Uh, λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω μετά τις θερινές διακοπές μας. Ελπίζω να περάσετε καλά και να έχετε προσέλθει εδώ ενθουσιώδης για να συνεχίσετε τη δουλειά. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, γιατί έχουμε αρκετά φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Δεν έχουμε ανακοινώσει του Προέδρου. Συνεχίζουμε με την έγκριση των πρακτικών. 18-19 Ιουνίου, 2 Ιουλίου, 9 Ιουλίου και 11-12 Ιουλίου. Επίση, ε, θέλουμε να εγκρίνουμε στο σημείο 4 το σχέδιο χρονοδιαγράμματο των συνεδριάσεων τη Επιτροπή για την περίοδο από Ιανουάριο έω Απρίλιο του 2019. Έχει συμφωνηθεί από του ε, συντονιστέ. Αν έχετε κάποιε αντιρρήσει πριν ε, από το τέλο τη σημερινή ημέρα, παρακαλώ να μα τι υποβάλλετε, γιατί πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα με το σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, έκθεση Γκαμπριέλ Μάτο για την ετήσια έκθεση τη Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017. Δεν θέλω ε, να του κλέψω τις ιδέες. Στην έκθεσή του όμως διαβάζω ότι μιλάει για την οικονομική κατάσταση και για το πρόγραμμα αγοράς τίτλων ε, και πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων και το ε, σύστημα ασφάλισης καταθέσεων. Θα δώσω όμως το λόγο στον εισηγητή για 5 λεπτά, μετά 4 λεπτά στους σκιώδεις εισηγητές και αν έχουμε το χρόνο και σύντομα διαδικασία κάτσου διάει. Κύριε Μάτο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Τεράστιος ο ενθουσιασμός του κοινού, όπως συνήθως συμβαίνει μετά το καλοκαίρι. Θα σε ευχαριστώ, εν πάση περιπτώσει. Θα μιλήσουμε για την οικονομική κατάσταση. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε στα πλαίσια της έκθεσης αυτής να ασχοληθούμε και με τα θέματα της νομισματικής πολιτικής, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το 2017 ήταν μια μεγάλη χρονιά ενισχύθηκε η ευρωπαϊκή οικονομία με τον ισχυρότερο ρυθμό της τα τελευταία δέκα χρόνια. Ε, υπάρχουν όμως μεγάλες διαφορές. Ε, εν πάση περιπτώσει τα θετικά οφείλονται και στις διαφθορτικές αλλαγές και στην νομισματική πολιτική. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat μας λέγουν ότι πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση οι προβλέψεις για το 2019 είναι γύρω στο 2% αύξηση της ε, δράστη του ΑΕΠ και θα φτάσουμε σε δεδομένα τα οποία θα έλεγα μας παραπέμπουν στην περίοδο που προηγήθηκε στις οικονομικής κρίσης. Αυτά επηρεάζουν θετικά και τον προϋπολογισμό βέβαια των ε, προϋπολογισμών της Ένωσης και της διαπραγματεύσεις για το Brexit και ο προστατευτισμός και ο λαϊκισμός εις βάρος της Ένωσης είναι στοιχεία τα οποία περιπλέκουν την κατάσταση και το βασικό είναι η οικονομική ανάπτυξη αυτή δεν έχει οδηγήσει σε πολλές δημιουργίες, ε, μάλλον σε δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας, δεν έχει υπάρξει μια πραγματική κοινωνική πολιτική που να παρομοιάζει με το τι συνέβαινε πριν από την κρίση. Απαιτείται λοιπόν γι' αυτό περισσότερη δράση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έτσι ώστε η, νομο, η πολιτική της ε, να μπορέσει να αποκαταστήσει την ε, πίστη ε, και τις πιστώσεις που πρέπει να προέρχονται από τον τραπεζικό τομέα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, κρατάει πάντα και γύρω στο 2% τον ε, <clears throat> πληθωρισμό και με τα μέτρα που έχουν ε, ληφθεί μέχρι τώρα δεν έχει ξεπεράσει παρασπάνια το 1,7%. Υπάρχει πάντα, υπήρξε μάλλον το πρόγραμμα αγορών ομολόγων. Είναι κάτι το οποίο έχει βοηθήσει να ισορροπήσει κάπως η κατάσταση και σε σχέση με το δημόσιο χρέος σε πάρα πολλές τις χώρες της Ευρώπης περνάμε σε μεγαλύτερη διαφάνεια και αντιμετωπίζουμε καλύτερα την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί με τις φούσκες στον τομέα των οικοδομών, σαν παράδειγμα σε ορισμένες χώρες τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν αντιμετωπιστεί γενικά θετικά, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ανίκανη να λύσει τα διαφορετικά προβλήματα των μεμονωμένων κρατών μελών. Τα ίδια τα κράτη-μέλη, ε, σε συνεργασία βέβαια με την ΕΚΤ, θα πρέπει να δουλέψουν στο διαρθρωτικό τομέα και ε, να βοηθήσουν έτσι συνολικά την Ευρωπαϊκή οικονομία, μία θα έλεγα πολιτική εκτατική στο τομέα της πίστοσης από πλευράς, το νομισματικό από πλευράς ευρωπαϊκής πολιτικής αφέ αυτής δεν είναι σε θέση να βοηθήσει αν δεν υπάρχουν μέτρα και μεταρρυθμίσεις διαφορετικές στα κράτη-μέλη που μόνον αυτές θα δημιουργήσουν τις συνθήκες που θα οδηγήσουν στη νομική ανάπτυξη τρία τελικά σημεία. Καταρχάς, η σημασία που έχουν οι διαπραγματεύσεις για το Brexit. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να είναι προπαρασκευασμένη για όλα τα πιθανά σενάρια. Ελπίζω να υπάρξει μια συμφωνία, ακόμα όμως και η δυνατότητα να προχωρήσουμε στο Brexit χωρίς συμφωνία είναι εδώ. Και ταυτόχρονα θα πρέπει και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αγορών και Κεφαλαίων θα βοηθήσει την καλύτερη μετάδοση των μέτρων της νομισματικής πολιτικής και θα ενισχύσει την εσωτερική αγορά. Και ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να έχει απόλυτη ελευθερία στη σχεδίαση της νομισματικής της πολιτικής σύμφωνα με τα δικά της κριτήρια αυτή νομίζω πρέπει να είναι η βάση όλων των διαπραγματευτών που έχουν πάρει μέρος μέχρι τώρα συζήτηση. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φερνάντες, εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα δεν είναι εδώ ο Γκλίντζο Μοριάνο και τον αντικαθιστώ. Έχω γραπτές σημειώσεις του τις οποίες μπορώ να διαβάσω. Η γενική του άποψη είναι ότι το σχέδιο έκθεσης είναι ισορροπημένο, αλλά έχει κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχήν, παίρνει το ρόλο της ΕΚΤ που υποστηρίζει ε, την οικονομική πολιτική, αλλά ε, χρειάζονται μέτρα οικονομικής και νομισματικής πολιτικής. Ε, δεύτερον, είναι σημαντικό να τονίζουμε τη σημασία του να υπάρχει ε, ε, ένας αντίστοιχος φορέας σε επίπεδο ευρωζώνης. Η Τρίτον, η ανεξαρτησία της ΕΚΤ είναι βασικός πυλώνας, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι εις βάρος της διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας. Και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το πλαίσιο αυτό. Τέταρτον, επίκυνται ε, εκλογές ε, για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ και για τον Πρόεδρό της και θα πρέπει να εξετάσουμε την σχετική εμπειρία ε, των υποψηφίων και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα για να υπάρχει και η σωστή ισορροπία μεταξύ γυναικών και ανδρών υποψηφίων. Ε, θέλουμε να συνεχίσει η ΕΚΤ να συνεισφέρει προς ε, τους στόχους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δημιουργηθούν συνέργειες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και επίσης, άλλο ένα σημείο, η ΕΚΤ θα πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση των πολιτικών κινδύνων που έχουν σχέση με τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Brexit. Έβδομο σημείο, στο πλαίσιο του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου, το Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί ε, το ρόλο της ΕΚΤ σε σχέση με τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελευταίο σημείο θέλουμε να διευκρινιστούν όλα όσα έχουν γίνει κατά τα χρόνια της κρίσης από την ΕΚΤ ε, με σκοπό ε, να έχουμε μια σαφή εικόνα και για τα περιουσιακά στοιχεία και τις πολιτικές της ΕΚΤ. Βέβαια, ο συνάδελφος ε, του οποίου διάβασα τις παρατηρήσεις θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με τον κύριο Μάτο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λούκ εκ μέρους του ECR. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς ο κύριος Λούνες δεν είναι εδώ σήμερα στην ανταλλαγή απόψε αυτή. Ζητά συγγνώμη διότι παρουσιάζει στην Επιτροπή Ίντα μια έκθεση του. Γι' αυτό και με παρακάλεσε να σας διαβάσω τα εξή. Καταρχάς ευχαριστεί τον εισηγητή για την ενδιαφέρουσα έκθεση. Η φετινή έκθεση δεν είναι μακροσκελής. Επικεντρώνεται σε βασικά ζητήματα που απασχολούν και εμάς ως ομάδα. Ε, ιδίως μας ε, ενδιαφέρει η επικέντρωση στην ε, κατάργηση του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων και την ε, σχετική μείωση του κινδύνου για τη δημιουργία οικονομικών, οικονομικής φούσκας. Επίσης, υπάρχουν, ε, ε, αναδεικνύονται και κάποιες ανισορροπίες ιδίως όσον αφορά τον πυλώνα 2. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιες ελλείψεις. Δυστυχώς η ανάκαμψη που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι ανεμική. Αν θέλουμε να επιστρέψουμε σε μια ισχυρή ανάκαμψη ε, και σε μεγαλύτερη δανειοδότηση χρειάζονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης θέλουμε να αναφέρουμε να αναφερθούμε στις αρνητικές επιπτώσεις που είχε το APP στους ε, ε, ε, ε, δανειολήπτες και τα νοικοκυριά. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τον συγγητή βεβαίω για αυτά τα θέματα. Εκ μέρους του Άλτη, κύριε Κρέντς, θέλετε να μιλήσετε. Όχι. Πολύ γρήγορα το πάμε. Δεν βλέπω κάποιον από τους πράσινους, ε, την ΚΟΕ, ή άλλες ομάδες. Επομένως, έχουμε λίγο χρόνο για διαδικασία Catch the, Eyes. Catch the Eye. Αν κάποιος θέλει να παρέμβει να τοποθετηθεί. Όχι. Α, ο κύριος Ροζάτη, παρακαλώ. Μία πρόταση θέλω να κάνω, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι μια σημαντική πολιτική εξέλιξη επίκειται. Η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει τα προγράμματα αγοράς περιουσιακών στοιχείων και αυτό θα πραγματοποιηθεί και στο πλαίσιο της αλλαγής που θα υπάρξει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ του χρόνου. Νομίζω ότι πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα για το πώς θέλουμε εμείς να εκτελεστεί αυτή η μετάβαση στην, ε, στην, την, την, ε, επάνωδο στην ομαλότητα στην νομισματική πολιτική και πώς αυτό θα θέλαμε να εκφράζεται και να προσανατολίζεται και μέσω της διοίκησης της ΕΚΤ μέσω της συνεργασίας με άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρούμε ότι πρέπει να, ε, θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί ε, ε, υπέρ της ανάπτυξης της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως. Το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων βεβαίως ήταν αμφιλεγόμενο οι επιπτώσεις αυτού και ο αντίκτυπός του έχει ασκηθεί σοβαρή κριτική γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει να αποσταλεί από την πλευρά μας ένα ισχυρό μήνυμα σε σχέση με αυτά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κάποιος άλλος, όχι. Να πω εγώ κάτι. Σκοπός μας και καθήκον μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι η ΕΚΤ θα μπορεί να κάνει τη δουλειά της, ακριβώς γιατί η νομισματική πολιτική μπορεί να προκαλέσει ε, μεγάλη δυσαρέσκεια σε πληθυσμιακές ομάδες ε, και σε ε, πολιτικούς χώρους. Θεωρώ ότι η ΕΚΤ πρέπει να έχει όλα τα εφόδια προκειμένου να υλοποιήσει την νομισματική πολιτική που χαράζει. Ο εισηγητή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συναδέλφους πήραν μέρος στη συζήτηση. Ε, συμμερίζομαι τις περισσότερες από τις παρατηρήσεις που έγιναν. Είναι προφανές ότι η έκθεση αυτή έχει σαν στόχο να βελτιωθεί η πρόταση που κάνω μάλλον να βελτιωθεί μέσω των προτάσεων και των τροπολογιών των συναδέλφων και να αποκτήσει ένα σωστό προσανατολισμό. Θα πρέπει να τα διευκρινίσουμε κάπως καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχει ένα θέμα θα ήθελα να πω ότι από μόνη της ε, είναι ένα θέμα αυτό η νομισματική πολιτική και η πολιτική στον τομέα των σχεδίασης των προϋπολογισμών από μόνη της από μόνες τους δεν ε, είναι σε θέση να βρουν λύσεις υπάρχει ανάγκη και από συνοδευτικές πολιτικές υπάρχει ανάγκη και από την εγγύηση που θα πρέπει να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την απόλυτη ανεξαρτησία της. Υπάρχει και το θέμα της λογικής των φύλων που θα πρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ και θα συνεχίσουμε την δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κλείσω θυμίζοντας ότι η προθεσμία είναι για την κατάθεση των τροπολογιών η 14η Σεπτεμβρίου. Η εξέταση θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου, θα ψηφίσουμε τον Νοέμβριο και στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου θα ψηφιστεί η έκθεση ΜΑΤΟ. Τώρα περνάω στο 6. Θα κάνουμε 5 λεπτά διάλειμμα γιατί περιμένουμε τον εισηγητή και θα ξεκινήσουμε πάλι σε, ε, ε στις 9.30. 5 λεπτά διάλειμμα λοιπόν.

So please let me go back to our agenda. Λοιπόν, να επανέλθουμε στην ημερησία διάταξη. Σημείο 6, έκθεση Μαυρίδη για τις οικονομικές πολιτικές της Ευρωζώνης. Εισαγωγικά θα ήθελα να πω ότι είναι μία από τις δύο συμβολές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξημείνου Άλλαξε ο εισηγητής, ο κύριος Μαυρίδης έχει αντικαταστήσει τον κύριο Μπαγιέ. Ήταν αρκετές οι τροπολογίες, 328 που κατατέθηκαν και που εξετάστηκαν για την έκθεση. Να δώσω το λόγο στον συγητή και στη συνέχεια στους κοιόδες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Και δεδομένου ότι είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε μετά το καλοκαίρι. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ όλους και να ευχηθώ να έχουμε μια αγώνιμη περίοδο τους επόμενους μήνες. Όπως είπατε, πράγματι ήταν αρκετές οι τροπολογίες, 328, που κατατέθηκαν. Και θεωρούμε πολύ σημαντικό την ε, έγκριση του εξής σημείου, που είναι και βασικό δική μας ανησυχία και που περιγράφεται και στις, στις ε, τροπολογίες μας. Πρώτον, περισσότερη ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή του ε, Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Εξαίρεση των δημόσιων επενδύσεων για την, ε, τον υπολογισμό του δημόσιου χρέους ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, ενσωμάτιση των εργασιακών και περιβαλλοντικών τον στους ε, στόχους για τη, για βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους του Παρισίου ώστε να λαμβάνονται υπόψη ε, στο, στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Καλύτερη ε, εξειδίκευση των συστάσεων αναχώρων. Τέταρτο, μεταρρυθμισμένο ευρωπαϊκό εξάμεινο με απότερο στόχο την ενίσχυση των, της ε, υλοποίησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα καθοδηγήσουν την κοινωνική και περιβαλλοντική μετάβαση και μεταρρύθμιση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Προώθηση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως σε κράτη-μέλη όπου η οικονομική κρίση είχε το μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο. Υποστήριξη της διαρθρωτικής χρηματοδότησης αντί της προτινόμενης μείωσης που προτείνει η Κομισιόν. Κατανομή των ευρωπαϊκών κονδύλιων υπό την αίρεση του ευρωπαϊκού εξαμήνου και, του, και της οικονομικής διακυβέρνησης είναι μια πολιτική που αντίκειται στην οικονομική ανάπτυξη. Η καταπολέμηση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στην Ευρωζώνη είναι εξαιρετικά σημαντική για την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Ο έλεγχος του άδικου χαρακτήρα των πρακτικών που εφαρμόζονται από τον τραπεζικό τομέα στις ε, συμβάσεις καταναλωτών πρέπει να καταπολεμηθεί και να υλοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Τέλος, η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης είναι σημαντικό στοιχείο, καθώς είναι βασικό στοιχείο μιας ε, εμβαθυμένης νομισματικής και οικονομικής ένωσης. Αμοιβεοποιημένο της έως το 2022 είναι ο στόχος μας. Κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να εντάξουμε στι συμβαστικέ τροπολογίε τι περισσότερε τροπολογίε που έχουν κατατεθεί. Και προσβλέπουμε σε μια γόνιμη και γνήσια συζήτηση, μια επικοδομητική συνεργασία στι συναντήσει των σκιωδών με όλε τι πολιτικέ ομάδε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα εισαγωγικά σα λόγια αυτά. Σκιώδη του ΕΛΚ είναι ο κύριο Φαντικάντελα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους. Είναι η πρώτη μας ε, συνάντηση μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Για την έκθεση αυτή βλέπω ότι παράλληλα με τα πολύ σημαντικά θέματα που συζητούνται υπάρχουν κάποια σημεία που δεν ε, περιλαμβάνονται στην ε, έκθεση και τα έχω σημειώσει και θα ήθελα να τα διατρέξουμε. Οι συστάσεις αναχώρα είναι το πρώτο. Το κόστος του πληθυσμού που γυράσκει είναι το δεύτερο και η αύξηση της παραγωγικότητας. Θα τα εξηγήσω όλα αυτά τα σημεία. Καταρχήν όταν μιλάμε για εργαλεία ανάπτυξης για την Ευρωζώνη, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε τους κανόνες για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη. Αυτά θα πρέπει να συμβαδίζουν με τα υπόλοιπα μέτρα. Θα πρέπει να εξετάζουμε την ανάπτυξη στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, όχι μόνο από πλευράς συντονιστικής. Πρέπει να έχουμε ε, υγιή δημοσιονομική κατάσταση. Κάτι το οποίο δεν αναφέρει η έκθεση, κατά τη γνώμη μου, είναι οι δυσκολίες στην ε, υλοποίηση. Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε. γιατί μόνο 9% των συστάσεων υλοποιούνται στην πράξη. Δεν υπάρχει λόγος να υποβάλλονται περαιτέρω συστάσεις αν δεν εφαρμόζονται οι συστάσεις οι οποίες ήδη υπάρχουν. Ε, όσον αφορά ε, τη γύρανση του πληθυσμού, είναι σημαντικό ε, να το συζητήσουμε γιατί είναι ένα βασικό πρόβλημα. Πρέπει να συζητήσουμε το θέμα των συντάξεων κλπ. Θέλουμε να έχουμε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και χρειαζόμαστε τις ε, σωστές δημοσιονομικές προβλέψεις για να έχουμε τις δημόσιες υπηρεσίες ε, που απαιτούμε. Ε, άλλο ένα σημείο έχω σχετικά με τις επενδύσεις. Η έκθεση μιλά για δημόσιες επενδύσεις, πράγμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε, αλλά παράλληλα να τονίσουμε και το ρόλο των ιδιωτικών επενδύσεων στην έκθεση. Είναι σημαντικό θέμα για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών και εδώ υπάρχει δυναμικό για τον τομέα αυτό. Τέλος, όταν μιλάμε για αύξηση μισθών, αυτό θα πρέπει να συνδυάζεται με την παραγωγικότητα. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και προσβλέπω στην συνεργασία σε μελλοντικές συναντήσεις των ε, σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε κάποιον από το ECR. Θέλετε το λόγο. Όχι. Καρολίνα Κτυγκαλ από το Άλντε. Τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Μαυρίδη που ανέλαβε την έκθεση αυτή και θα συνεργαστούμε στενά κατά τους επόμενους μήνες είδα τις διάφορες τροπολογίες που υπέβαλαν οι συνάδελφοι και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ καλή βάση για τη μελλοντική μας συζήτηση. Με τις συστάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη, στόχος είναι η σύγκληση των εθνικών οικονομιών και θα πρέπει να φροντίσουμε να παρακολουθούμε τις σχέσεις με την οικονομική κρίση και την ανάκαμψη. Σήμερα φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει η ανάκαμψη και θα πρέπει να συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή και να γίνουν πιο συγκεκριμένες οι διάφορες μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται. Θεωρώ απογοητευτικό το ότι κάποιες συστάσεις της Επιτροπής δεν τηρούνται. Ε, και βέβαια γνωρίζουν τα κράτη-μέλη της συστάσεις, αλλά δεν είναι έτοιμα να τις εφαρμόσουν και να τις εντάξουν στην στρατηγική τους. Είναι λυπηρό και είναι και ανεύθυνη στάση. Ορισμένοι συνάδελφοι ανέφεραν ε, τους δημοσιονομικούς κανόνες ε, και ε, το πόσο ευέλικτη θα μπορούσε να είναι και όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας μας χρειάζεται μια ευελιξία αλλά η αγορά εγγυάται την απασχόληση και όχι ο δημόσιος τομέας αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε τη δημοσιονομική εξυγίανση και να ε, φροντίσουμε ώστε να συνεχιστεί η ανάκαμψη. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο υποβάλαμε και εμείς τροπολογίες για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί με στόχο την σταθεροποίηση των οικονομιών. Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να συνεχίσουν προς την επιθυμητή κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ένωση Κεφαλή Αγορών. Θα πρέπει να παίξει ο καθένας το ρόλο του και εμείς ε, ε, ως κοιόδης ε, εισηγητές, σε συνεργασία με τον εισηγητή, θα συνεχίσουμε την επεξεργασία της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Ο κύριος Στάσον από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαυρίδη και τον κύριο Μπαγιέ για το σχέδιο έκθεσης που συζητούμε. Προσβλέπω σε συνεργασία με τους υπόλοιπους σκιώδεις για να καταλήξουμε σε μια θετική έκθεση. Νομίζω ότι το κείμενο αποτελεί θετική βάση για το διάλογο. Υπάρχει καλή διάγνωση της οικονομικής κατάστασης και επικεντρωνόμαστε σε βασικά ζητήματα δίκη φορολόγηση, μείωση ανεργίας και ενίσχυση των ε, μεταρρυθμίσεων. Επίσης αναγνωρίζει τις ε, ανισότητες και ανισορροπίες ε, στις ευρωπαϊκές οικονομίες, ιδίως στο υπερβολικό πλεόνασμα ορισμένων χωρών. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει επαρκής κριτική σε κάποιες ευρωπαϊκές πολιτικές. Η που έχει προωθηθεί από την Κομισιόν δεν κατάφερε να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση, ούτε να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο των πολιτών, να προστατεύσει το περιβάλλον και να εξασφαλίσει κάποια ελάχιστα πρότυπα στα κράτη-μέλη. Θεωρούμε ότι η κοινωνική και περιβαλλοντική στόχοι περιλαμβανομένων των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και των Παρισίων πρέπει να αποτελέσουν στόχο και της των πολιτικών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τροπολογίες μας ε, επικεντρώνονται στην ανάγκη μείωσης των ανισοτήτων και της προώθηση μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης για την ε, φορολόγηση ε, υποβάλαμε τροπολογία όπου ε, επενούμε την Κομισιόν για την προτάσή της να καταπολεμηθεί η επιθετική φορολογική πολιτική ε, στην 110 καλούμε την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να ε, εξασφαλίσουν και να προστατεύσουν ε, τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις που έχουν υπονομευθεί από κάποιες συστάσεις αναχώρα. Επίσης σημαντικό είναι για εμάς να ενισχυθεί και να εξασφαλιστεί η μετάβαση στην κυκλική οικονομία και μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Ε, επίσης, σημαντικό είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς σε κάποια κράτη-μέλη. Η διαφθορά έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και για το επιχειρηματικό περιβάλλον. Η 328 μας, ε, η τροπολογία μας καλεί να ε, τεθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι σε αυτό το θέμα. Και τέλος, να τονίσω και εγώ αυτό που είπε ο εισηγητής, ότι χρειάζεται πολιτική βούληση για να προχωρήσει η Τραπεζική Ένωση και να ξεμπλοκαριστεί το έντις, ε, κάτι που είναι τελείως απαράδεκτο αυτή τη στιγμή, το γεγονός ότι είναι μπλοκαρισμένο. Αλλά, όπως είπα, προσβλέπουμε και στη συνεργασία με τους υπόλοιπους σκιώδεις για να καταλήξουμε σε ένα θετικό κείμενο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Η θέση μας σχετικά με το ευρώ είναι σαφής. Εμείς είμαστε κατά του ευρώ, είμαστε κατά των κανόνων ε, του ευρώ, είμαστε κατά της, ε, του προσανατολισμού και είμαστε κατά και των συστάσεων αναχώρα. Το ευρώ δεν έχει προσφέρει τίποτα, δεν έχει προσφέρει σταθερότητα, δεν έχουμε καταστεί αποτελεσματική οικονομικά, δεν έχουμε δει καμία μορφή αλληλεγγύης η εφαρμογή των κανόνων της ζώνης ευρώ και στη δική μου χώρα, την Πορτογαλία, έχει λειτουργήσει προκυκλικά έχει οδηγήσει στην οικονομική κατάρρευση και στην απώλεια οικονομικής ανεξαρτησίας. Χάσαμε όλες τις στρατηγικές επιχειρήσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στον τομέα των μεταφορών, όλα ελέγχονται από το διεθνές κεφάλαιο όλες οι υπηρεσίες κοινή ωφέλεια λειτουργούν πολύ λιγότερο ε, ικανοποιητικά λόγω της έλλειψης επενδύσεων ε, των τελευταίων ε, ετών. Ευτυχώς στην Πορτογαλία έχει υπάρξει μια πολιτική αλλαγή από το 2015 και μετά και έτσι καταφέραμε να απαλλαγούμε από πολλά από τα μέτρα τα οποία επέβαλε η Τρόικα και τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι αντίθετα με τις συστάσεις αναχώρα. Εμείς μειώσαμε τη φοροσλόγηση της εργασίας, εμείς μειώσαμε τους ρυθμούς ιδιωτικοποίησης και αυτά όλα βοήθησαν την οικονομία, μας λέγανε ότι θα βουλιάξουμε, έγινε ακριβώς το αντίθετο και γι' αυτό τα μέτρα λιτότητας που θέλουν να μας επιβάλλουν είναι η κακή συνταγή για τις περισσότερες χώρες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει η δυνατότητα στις χώρες οι οποίες βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση μέσα στη ζώνη ευρώ να μπορούν με ε, τακτό τρόπο να εγκαταλείπουν τη ζώνη ευρώ διασώζοντας την ανεξαρτησία τους. Σας ευχαριστώ. Από το EFTD υπάρχει κάποιος, από το ENF. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Catch the Eye. Θα ήθελε κάποιος το λόγο. Δεν θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Θα επανέλθω λοιπόν στον εισηγητή μας. Κύριε Μαυρίδη, αν θέλετε μπορείτε να κλείσετε τη συζήτηση. Νομίζω ότι υπόθηκαν όσα έπρεπε να υποθούν. Σημειώνουμε ε, ότι θα υπάρξει θετικός διάλογος και συζήτηση και προσβλέπουμε σε αυτή τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ελπίζουμε και εμείς ε, ότι θα ακολουθήσει αυτή η επικοδομητική συζήτηση. Στις 9 Οκτωβρίου ε, θα ακολουθήσει η ψηφοφορία στην Επιτροπή Οικών και θα συζητηθεί στη δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου. δεν βλέπω τον εισηγητή μας για το επόμενο θέμα. Βλέπω τους μισούς εισηγητές, το 50% τον κύριο Τάγκ. Μάλλον, ο κύριος Τάγκ είναι ο ένας που απουσιάζει, είναι το 50% που απουσιάζει και μόλις εμφανιστεί θα συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ψηφιακή ε, οικονομία. Ευχαριστώ. Grande

Να συνεχίσουμε. Έχουμε μία ώρα για να συζητήσουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Δύο προτάσεις που σχετίζονται με την ε, φορολόγηση των εταιριών με σημαντική ψηφιακή παρουσία. Οι βασικές έννοιες που βρίσκονται σε αυτούς τους φακέλους είναι πρώτον η ε, ψηφιακή παρουσία και η Κομισιόν το Μάρτιο ε, πρότεινε κάποια ε, ενδιάμεσα μέτρα για το πώς θα χειριστούμε αυτήν την ενοποιημένη βάση φορολόγησης σε σχέση με την σημαντική ψηφιακή παρουσία και προτείνονται και κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που είχε προτείνει άλλωστε και το, το Κοινοβούλιο όσον αφορά την CCTB και την CCCTB. Έχουμε λοιπόν 60 λεπτά για να συζητήσουμε αυτά τα δύο θέματα και γι' αυτό έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε 10 λεπτά στον κάθε εισηγητή. Πρώτα στον κύριο ε, Ροζάτη που είναι υπεύθυνο για το θέμα των μακροπρόθεσμων λύσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον πακέτο προτάσεων. Είναι ένα που το έχουμε συζητήσει ήδη εδώ στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των ε, επιτροπών τάξε 1, 2 και πάνω και αποτέλεσε θέμα βεβαίως και των συζητήσεων που έγιναν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρωτοβουλία της Κομισιόν που υπέβαλε αυτές τις δύο νομοθετικές προτάσεις αντικοτοπτρίζει την ανησυχία ότι οι ψηφιακές επιχειρήσεις διαφέρουν από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις όσον αφορά τις εφορολογικές τους υποχρεώσεις. Οι ψηφιακές εταιρείε λειτουργούν με βάση ένα τελείως διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο σε σχέση με τις ε, Παραδοσιακέ εταιρείε με τη φυσική παρουσία τους. Όπου ένα από τα βασικά στοιχεία του των παραδοσιακών εταιρεών, ήταν ότι ε, παρήχαν υπηρεσίες και προϊόντα μέσω της φυσικής τους παρουσίας απέναντι στους καταναλωτές. Κάτι που ήταν πολύ εύκολο και στην, ε, ε, για τη δουλειά των φορολογικών αρχών. Στις ψηφιακές εταιρείε υπάρχει μια διάκριση μεταξύ αυτών των δύο χαρακτηριστικών. Δηλαδή, μια εταιρεία μπορεί να παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς να έχει καμία φυσική παρουσία σε κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα η, τα αγαθά που ε, προσφέρει είναι άειλα και που εξορισμού είναι πολύ είναι πολύ δύσκολο να, τα, να αποτιμήσει κανείς την αξία τους. Και επιπλέον οι ψηφιακές εταιρείες βασίζονται σε, αυτήν την, σε αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο τύπο ε, παραγωγής αξίας που είναι η συμμετοχή των χρηστών. Όσο περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν ένα δίκτυο ή επισκέπτονται μια ιστοσελίδα, τόσο μεγαλύτερη ε, ε, γίνεται η αξία αυτή τη υπηρεσία. Υπάρχει λοιπόν μια διάδραση μεταξύ τη εταιρεία και των χρηστών. Όσο περισσότερο χρησιμοποιούν οι χρήστε μια συγκεκριμένη υπηρεσία, τόσο περισσότερο αυξάνεται η αξία αυτή τη υπηρεσία. Αυτό είναι ένα στοιχείο που διακρίνει και που καθιστά μοναδικέ τι ψηφιακέ εταιρείε. Και στο πλαίσιο της πρότασης που συζητούμε αντιμετωπίζουμε ε, σημαντικότατα προβλήματα εμείς και οι φορολογικέ αρχές, δηλαδή, ω προ το πώς θα φορολογηθούν αυτές οι δραστηριότητες. Υπάρχει μια ε, απόκληση μεταξύ της πηγής και της ε, μόνιμης κατοικίας, ε, για παράδειγμα. Ε, αλλού, σε μια χώρα μπορεί να παρέχεται ε, μια υπηρεσία και η έδρα της εταιρείας που παρέχει την υπηρεσία αυτή βρίσκεται σε άλλη χώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να, μπορεί, να μπορέσει κανείς να τα συνδέσει αυτά και να καθορίσει ποιο τμήμα της αξίας της υπηρεσίας αυτής θα πρέπει να ε, ε φορολογηθεί σε ποια χώρα. Όλα αυτά τα ζητήματα μας απασχολούν. Βεβαίως συμφωνούμε όλοι ότι κάτι πρέπει να γίνει με τις ψηφιακές εταιρείε και αυτό είναι και το συμπέρασμα στο οποίο έχουμε καταλήξει ε, ε, και στο οποίο κατέληξε και ο ΣΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν πάρα πολλές γνωμοδοτήσεις, απόψεις ε, που ε, αναφέρουν ότι η φορολόγηση των ψηφιακών επιχειρήσεων, των ψηφιακών εταιρεών δεν είναι δίκαιη. Ιδίως των πολύ μεγάλων εταιρεών αυτών και κάτι πρέπει να γίνει. Επί της αρχής η Κομισιόν προσπαθεί να απαντήσει στα εξής ερωτήματα. Πρώτον, δηλώνει ότι θέλει να φορολογήσει τις ψηφιακές εταιρείες δηλώνουν... Αλλά το, το ερώτημα είναι ε, με ποιον τρόπο. Το δεύτερο ερώτημα είναι πού θα φορολογηθούν οι ψηφιακές εταιρείε όταν παρέχουν υπηρεσίες σε διάφορες χώρες. Και δεδομένου ότι πολλές από αυτές τις υπηρεσίες ε, είναι και ε, διασυνοριακές. Και βεβαίως τρίτο ερώτημα πόσο να φορολογηθούν. Οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες και οι περισσότεροι πολίτες συμφωνούν ότι κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά δυστυχώς εκεί τελειώνει και η συμφωνία γιατί κάθε άλλη επιλογή που προτείνεται από τον ΟΣΑ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προκαλεί διχογνωμία και δεν μπορεί να προχωρήσει η συζήτηση. Ε, υπήρξε λοιπόν η ιδέα ότι Α, η καλύτερη δυνατή λύση θα ήταν μια διεθνής λύση. Λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα το, της παροχής των ψηφιακών υπηρεσιών. Αλλά για να επιτευχθεί διεθνή συμφωνία σε επίπεδο όσα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ούτε προβλέπεται να γίνει κάτι τέτοιο στο άμεσο μέλλον. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την πρωτοβουλία και να προτείνει μια λύση η οποία ενδεχομένως δεν θα είναι η μακροπρόθεσμη διαρθρωτική λύση ε, που θα διαρκέσει για πάντα, αλλά τουλάχιστον θα μπορέσει να απαντήσει σε ορισμένα από τα προβλήματα που έχουν ανακύψει ε, και μια τέτοια κίνηση θα ανοίξει το δρόμο για να ξεκινήσει η συζήτηση και με άλλες χώρες. Υπάρχει, λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν δύο εκθέσεις. Η μία που αφορά την, τη διαρθρωτική, την ε, οριστική λύση που θα δοθεί στο θέμα αυτό και υπάρχει και η άλλη έκθεση που θα συζητήσουμε αργότερα για τα ενδιάμεσα μέτρα που θα ληφθούν. Η πρόταση για την διαρθρωτική λύση βασίζεται στην πρόταση να οριστεί αυτός ο όρος της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας. Ένας τέτοιος ορισμός θα έδινε τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να καθορίσουν πού ακριβώς παράγεται η αξία. Η σημαντική ψηφιακή παρουσία δεν ταυτίζεται με την φυσική παρουσία, μπορεί και να ταυτίζονται ή να επικαλύπτονται, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το ότι λέμε ότι μια εταιρεία που έχει την έδρα της στη ΣΥΠΑ μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της στη Γαλλία χωρίς να έχει καθόλου φυσική παρουσία στη Γαλλία, αλλά επειδή παρέχει τις υπηρεσίες της στην Γαλλία θα πρέπει με κάποιον τρόπο να προσδιοριστεί η ε, σημαντική αυτή ψηφιακή παρουσία της, ακόμα και αν δεν υπάρχει φυσική παρουσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προτείνει αυτή η σημαντική ψηφιακή ε, παρουσία να βασίζεται σε τρία κριτήρια. Πρώτον, όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των συμβάσεων και τον αριθμό των χρηστών. Τρία κριτήρια. Το μόνο ερώτημα που έχω να θέσω εγώ είναι γιατί ορίστηκαν αυτοί οι δείκτες. 7 ε, εκατομμύρια για το κύκλο ε, εργασιών, 100.000 χρήστες και 3.000 συμβάσεις. Με ποιον ακριβώς τρόπο και για ποιον ακριβώς λόγο ε, επιλέχθηκαν αυτά τα όρια. Με ποια λογική. Και αν πράγματι μας βοηθούν αυτοί οι δείκτες για να καλύψουμε όλες τις εταιρείε με σημαντική ψηφιακή παρουσία. Διότι έχει αποδειχθεί ότι σε κάποιες πολύ μικρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να μην πληρούνται, να μην, να μην πληρούνται τα κριτήρια αυτά. Αν στόχος μας είναι να ε, θέσουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας τις μεγάλες εταιρείες, τότε εντάξει. Αλλά θεωρώ ότι είναι, θα ήταν σωστό και δίκαιο ε, να θέσουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας όλες τις εταιρείες με ψηφιακή παρουσία. Αυτά ως προς την διαρθρωτική λύση και όπως καταλαβαίνετε αν καταλήξουμε σε ορισμό της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας από εκεί και πέρα βεβαίως ε, η Επιτροπή ε, προτείνει και συγκεκριμένους τρόπους ε, για την ε, φορολόγηση ή για την εκτίμηση των ψηφιακών δραστηριοτήτων, τον προσδιορισμό της αξίας τους δηλαδή, κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα αργότερα στα κράτη-μέλη και στις φορολογικές τους αρχές να εντάξουν τις εταιρείες αυτές στην ενοποιημένη βάση φορολόγησης εταιρεών. Αυτή είναι η διαθροτική λύση, έτσι με έναν πολύ ευσύνοτο τρόπο σας τα παρουσίασα τα ερωτήματα που έχουμε να θέσουμε εμείς στις όσον αφορά τις προτάσεις αυτές, σε αυτό το πολύ πρώιμο στάδιο των συζητήσεων, ε, είναι ε, πολλά, αλλά εγώ σήμερα θα επικεντρωθώ μόνο σε δύο-τρία. Αναφέρθηκα ήδη στο ζήτημα του προσδιορισμού αυτών των συγκριτικών δικτών που έχουν τεθεί. Κάτι άλλο που με εξέπληξε όταν ε, διάβασα το έγγραφο είναι ότι ο ορισμός των ψηφιακών υπηρεσιών είναι αρκετά ασαφής. Και μάλιστα ανοίγει, αφήνει ανοιχτή την πόρτα και σε παρεξηγήσεις. Υπάρχουν ε, υπηρεσίες που χρησιμοποιούν δίκτυα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν μέσα πληρωμής. Αυτές οι τελευταίες εταιρείε δεν καλύπτονται από την οδηγία, την προτινόμενη. Το ερώτημά μου λοιπόν προς τους εκπροσώπους της Κομισιόν είναι πώς μπορεί να γίνει η διάκριση μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών εταιρεών Και για ποιο λόγο βεβαίως να μας απαντήσουν εντάσσεται η πρώτη κατηγορία στην οδηγία και η άλλη όχι. Το τρίτο πράγμα που θέλω να θέσω είναι το εξή. Έχω κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά τον, την πρακτική εφαρμογή, εφαρμοσιμότητα καλύτερα, του συστήματος. Κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί νέα υπηρεσία να δημιουργηθεί σε κάθε κράτος μέλος. Αλλά θα χρειαστούν και ε, μεθοδολογίες και ε, τεχνικός και τεχνικές δυνατότητες εν γέννη προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι ψηφιακές εταιρείες ε, ακολουθούν και τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις που να προτείνονται και γι' αυτό δεν έχω καταλάβει, ε, μάλλον έχω τις αμφιβολίες μου ότι θα μπορέσουμε πραγματικά να καθορίσουμε με απόλυτη βεβαιότητα ε, ε, ότι η οδηγία θα εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες και ότι δεν θα ξεφεύγουν κάποιες από τις δραστηριότητες στο, στην ψηφιακή σφαίρα με διάφορες προφάσεις. Τέλος, Όσον αφορά το, το ζήτημα της συνολικής συμφωνίας, ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο απλά γνωμοδοτεί. Από τη μελέτη αντικτύπου γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιθέσεις και διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών στα ζητήματα αυτά. Θα ήταν θετικό να μάθουμε πόσο μεγάλε είναι αυτέ οι διαφωνίε. Υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι υπέρ τη πρότασης, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες χώρες που αντιτίθενται στην πρόταση αυτή γενικά. Καθώς δεν θέλουν καμία νομοθετική ρύθμιση του θέματος αυτού, ε, φέρουν διάφορες προφάσεις όπως είναι η αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης, διοικητικό κόστος κτλ. Θα ήταν ε, θετικό λοιπόν να γνωρίζουμε ποιες είναι οι πιθανότητες το Συμβούλιο στο επόμενο διάστημα να καταλήξει σε συμφωνία. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο και στον κύριο Χορτάν για... που είναι εισηγητής για το δεύτερο θέμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω μετά από αυτό το μεγάλο διάλειμμα. Ελπίζω να περάσατε όλοι καλά. Έχουμε μπροστά μας ένα φάκελο τον οποίο έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για τη φορολογία αυτή. Και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει μια προφανέστατη αδικία εδώ. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις πληρώνουν πολύ λιγότερο φόρο από τις μικρόμεσες και υπάρχουν και τρομακτικές διαφορές ανάμεσα στις πολυεθνικές η Google, το Facebook, οι πλατφόρμες αυτές δεν πληρώνουν το φόρο που θα έπρεπε. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό είναι κάτι το άδικο και είναι κάτι το οποίο επηρεάζει το φορολογικό ήθος αν θέλετε. Γιατί κάποιος να πληρώνει περισσότερα από κάποιον άλλον. Αλλά ακόμα και αν δεν το βλέπει κανείς ε, σαν κάτι το άδικο είναι κάτι το αναποτελεσματικό δεν δημιουργείται μία θα έλεγα δίκαιη κατανομή της φορολογίας και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα κοινό τρόπο να κάνουμε κάποιες προτάσεις στον τομέα της φορολογίας των επιχειρήσεων. Είτε θεωρείτε ότι είναι άδικο, είτε θεωρείτε ότι είναι αποτελεσματικό, πρέπει να το διορθώσουμε προτείνονται κάποιες λύσεις οι οποίες είναι λίγο δύσπεπτες θα έλεγα. Καταρχάς η πρώτη λύση είναι το να μην κάνουμε τίποτα. Αυτό το πιστεύουν χώρες όπως η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. Το να μην κάνουμε τίποτα στην ουσία η αναποτελεσματικότητα και η αδικία θα συνεχιστούν σε τρομακτική κλίμακα και νομίζω ότι αυτή δεν μπορεί να είναι η επιλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια πιο ελκυστική αλλά παρόλα αυτά δύσκολη λύση είναι να περιμένουμε να υπάρξει λύση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Google είπε ότι ναι, να πληρώνουμε φόρο αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Προφανώς το λέει αυτό γιατί ξέρει ότι θα πρέπει να περιμένει αιώνες για να το πετύχουμε αυτό. Το λέει εύκολα λοιπόν, αλλά δεν ισχύει. Συνεπώς λοιπόν δεν νομίζω ότι είναι μία λύση το να περιμένουμε τον ΩΣΑ. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό φόρουμ ο ΩΣΑ, αλλά νομίζω ότι απαιτείται μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για να αντιμετωπιστεί το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση απέναντι στους εκλογείς μας να αντιμετωπίσουμε τις αναποτελεσματικότητες της φορολογίας. Θα πρέπει να πάρουμε πρωτοποριακό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και να δημιουργήσουμε τα νέα επίπεδα αναφοράς για τον 21ο αιώνα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη δείξει την σωστή κατεύθυνση, υπήρξε στήριξη για το CCCTB ήμουν πάλι εισηγητή και ήταν επίσης και ο Λαμασούρ κύριος εισηγητής. Αυτό προκάλεσε μια βασική αλλαγή στην φορολογία των επιχειρήσεων γιατί δεν αναζητούμε ε, με τον τρόπο που το κάναμε αυτό τα κέρδη και σε επίπεδο ψηφιακών ε, ε, δραστηριοτήτων και σε επίπεδο σωστής φορολόγησης των κερδών εκεί όπου παράγονται. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι έτσι μόνο θα μπορέσουμε να αναζητήσουμε την βελτίωση της κατάστασης και να τύχουμε της υποστήριξης της πλειοψηφίας. Έδωσα λοιπόν κάποια πρώτα θα έλεγα επιχειρήματα ο φόρος κύκλου εργασιών είναι θα έλεγα κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν δυνατότητα. Έτσι μόνο η Ευρώπη θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την αδικία και την αναποτελεσματικότητα του ισχύοντος συστήματος και έτσι μόνο θα πιέσουμε και τον ΟΣΑ και τις άλλες χώρες. Λοιπόν, το DST, το Digital Services Turnover Tax θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με πιο διαφορετικό τρόπο από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα κάνει. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θεωρώ ότι είναι ένα μέσο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και το οποίο θα επιτρέψει περαιτέρω αλλαγές. Μια ένα ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε την διάκριση ανάμεσα σε αυτά τα οποία υπάρχουν ε, στην ε, πρόταση για την ενιαία φορολογική βάση των επιχειρήσεων και στο πεδίο στο οποίο παράγεται, ε, δημιουργείται αν θέλετε η συγκεκριμένη παραγωγή ψηφιακού τύπου. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει την επιβολή φορολογία σε ένα τμήμα των επιχειρήσεων και όχι μόνο στο σύνολό τους. Αλλά στα πλαίσια του CCTB, ότι ο φόρος τον οποίο πληρώνεις εξαρτάται από το που παράγεις και εξαρτάται επίσης και από το που γενικά κερδίζεις, από που συλλέγεις τα περισσότερα κέρδη σου. Συνεπώς λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει και αυτό να το εξετάσουμε γιατί η μακροπρόθεσμα σίγουρα θα μπορέσει να μας προσφέρει κάποιες λύσεις. Τώρα κάποια επιμέρους θέματα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στα πλαίσια του DST 3% ε, επί του κύκλου εργασιών. Αν δει κανεί τα δισεκατομμύρια τα οποία βγάζουν οι ψηφιακέ πλατφόρμες, ο Τζεφ Μπέζος είναι ο, ο, πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο και τον ακολουθεί ο Τσούκεμπεργκ και γι' αυτό το 3% είναι πραγματικά χαμηλό ενώ το 5% δεν είναι υπερβολικό. Γιατί να μείνουμε στο 3% μόνο και γιατί επίσης να μην αποφασίσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στις χώρες μας να επιβάλλουν το επίπεδο το οποίο επιθυμούν ακόμα και υψηλότερο αν αυτές το θέλουν. Συνεπώς λοιπόν δεν είναι υψηλός ο φόρος αυτός λόγω των υψηλών κερδών που ε, προσπορίζονται οι μεγάλες αυτές επιχειρήσεις. Νομίζω ότι η χρηματιστηριακή αξία των μεγάλων επιχειρήσεων δείχνουν ότι οι πρώτες επιχειρήσεις στον κόσμο είναι ε, το Facebook, ε, η Amazon, η Microsoft και η Apple. Συνεπώς λοιπόν δεν κινδυνεύουν από υπερβολική φορολογία. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει υψηλό επίπεδο επιβολής, θα πρέπει να είναι ε, ταυτόχρονα κοινό ε, και επίσης θα πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να φορολογηθεί και η πώληση δεδομένων. Νομίζω ότι ε, προφανώς και θα πρέπει να φορολογηθεί η πώληση των δεδομένων των προσωπικών γιατί αλλιώς κάποιες μεταφορές δεδομένων ανάμεσα σε επιχειρήσεις θα διαφεύγουν της φορολογίας ιδιαίτερα όταν γίνεται στο εσωτερικό των ομίλων, ε, θα διαφεύγουν εντελώς. Συνεπώς λοιπόν είναι σαφές ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο παράγει αξία και η πώληση δεδομένων είναι σαφές ότι θα πρέπει να φορολογηθεί γιατί δημιουργεί κέρδη και το συζητάμε τώρα το θέμα γενικά το φορολογικό σε σχέση και με το τι κάνουν με τα δεδομένα μας οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Τώρα για το τελευταίο λεπτό της παρέμβασής μου για την ε, μόνιμη εγκατάσταση, την μόνιμη έδρα είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί ε, στο Κοινοβούλιο εδώ και ένα χρόνο. Έχει υπάρξει μια απόφαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν και είναι μια λογική θα έλεγα προέκταση της, ε, του καθορισμού της ε, ψηφιακής παρουσίας όχι μόνο στα πλαίσια του CCTB αλλά και γενικότερα των, των, των φόρου επιχειρήσεων. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά στην υπεξεργασία των θέσεων εδώ. Είναι δύσκολο το θέμα και θα το εξετάσουμε εκ νέου. Βλέπω ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνει κάποια ανώτατα όρια, τα οποία μερικές φορές είναι υψηλότερα από αυτά που είχαμε προτείνει. Νομίζω ότι η σύλληψη αυτή λοιπόν αντικατοπτρίζει σωστά στοιχεία που προέρχονται όχι μόνο α στα πλαίσια του ε, κοινού πεδίου επιβολής ε, ε, των φόρων επιχειρήσεων αλλά και των εθνικών ρυθμίσεων. Εφόσον υπάρχουν κέρδη πρέπει να δούμε ακριβώς πώς μπορούν να φορολογηθούν, πώς μπορεί να κατανεμηθούν τα κέρδη αυτά και δεν καταλαβαίνω στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί δεν γίνονται πιο συγκεκριμένες προτάσεις και στα πλαίσια του CCTB των στοιχείων που παίρνουμε για τις πωλήσει, για το προσωπικό, για το εργατικό δυναμικό μάλλον. Έχουμε λύσει κάποια θέματα με το CCTB στον τομέα σαν παράδειγμα της ε, πνευμανικής ιδιοκτησίας. Και γιατί να επανερχόμεθα εξ αρχής λες και δεν έχουμε κάνει ε, κάτι. Πρέπει λοιπόν η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να δούμε ακριβώς πώς κατανέμονται τα κέρδη, πώς διαιρούνται τα κέρδη ανάμεσα στις επιχειρήσεις ενός ομίλου για να μπορέσουμε να, τις να τα Και θα πρέπει να δούμε πώς θα αναθεωρήσουμε εν περιπτώσει και θα μεταρρυθμίσουμε τον φόρο των επιχειρήσεων έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 21ου αιώνα υπάρχουν τεράστιες αναποτελεσματικότητες, υπάρχουν τεράστια επίπεδα αδικίας και έχουμε τεράστιες επιχειρήσεις, γιγαντιές επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν φόρους και θα πρέπει να δώσουμε εξηγήσει για την κατάσταση αυτή στις επερχόμενες εκλογές. Ευχαριστώ τον Τάγκ. Πριν περάσουμε στους Κιώδης να πω ότι έχουμε και ένα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η εκπρόσωπος ε, μπορεί να πάρει το λόγο εφόσον το επιθυμεί αλλά πριν γίνει αυτό να ακούσουμε παρακαλώ τους Σκιώδης μετά το Catch the Eye και μετά θα δώσουμε το λόγο ε, στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Τάγκ έχει ήδη εκφραστεί λοιπόν. Θα δώσω το λόγο στον Μάτο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σκιώδης για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και όλοι θα συμφωνήσουμε να πούμε ότι είναι από τις πιο σημαντικέ πολιτικές που απασχολούν τα ευρωπαϊκά όργανα και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα σταθερό και σύγχρονο φορολογικό σύστημα είναι θα έλεγα καθοριστικό για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων από την οποία θα ωφεληθούν εκατομμύρια Ευρωπαίων. Βλέπουμε ότι οι ψηφιακές επιχειρήσεις αναπτύσσονται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από το σύνολο της οικονομίας και μετασχηματίζουν τον τρόπο ε, διάδρασης ε, των πολιτών και προσφέρουν πάρα πολλά στις, ε, στην κοινωνία. Ο συσχετισμός λοιπόν της φορολογίας με τις ψηφιακές τεχνολογίες ε, δημιουργούν νέες ευκαιρίες, προσφέρουν νέες λύσεις και διευκολύνουν την συνεργασία ανάμεσα στις φορολογικές αρχές. Και νομίζω ότι καταπολεμούν, υπάρχουν μέσα και για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Λοιπόν, ε, βλέπουμε πώς ακριβώς δημιουργείται το πρόβλημα σήμερα, περιγράφεται το πρόβλημα σήμερα στα πλαίσια της ψηφιακής παραγωγής. Ο πεπαλαιωμένος χαρακτήρας των φορολογικών συστημάτων έχει οδηγήσει ε, στη μείωση των ε, εσόδων και στην μείωση γενικά της σημασίας της φορολογίας. Το να μιλάμε για τη φυσική παρουσία επιχειρήσεων σε έναν χώρο, σε μία χώρα μάλλον, δεν έχει μεγάλη σημασία γιατί ξέρουμε ότι η ψηφιακή παραγωγή δεν γίνεται. Πάντως σε διεθνές επίπεδο υπάρχει μια προϊούσα θα έλεγα αναγνώριση της ανάγκης να υπάρξει ένα νέο φορολογικό μέτρο και σύστημα το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες που έχει η ψηφιοποίηση της οικονομίας και εδώ παραπέμπουμε και στα πλαίσια των ε, εργασιών του ΟΣΑ ε, και στα πλαίσια των ε, μεγάλων ομάδων συνεργασιών των χωρών νομίζω ότι έχουν εντοπιστεί κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν ποιες είναι οι χώρες που θέλουν να εισάγουν έστω και μεμονωμένα μεταβατικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί ένα φορολογικό πρόβλημα το οποίο δημιουργείται από την ψηφιοποίηση της οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα προσωρινό πακέτο και έχει προτείνει και κάποιες προτάσεις για μακροπρόθεσμες λύσεις ε, είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς καμία αμφιβολία πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας αυτής. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να συζητήσουμε, πρέπει να δούμε ποια είναι τα στοιχεία, οι αριθμοί, τα ποσοστά, αλλά είναι σαφές ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στη συζήτηση του πακέτου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τίθενται λοιπόν τα θέματα. Πρέπει να ακούσουμε επίσης και τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων για να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος αυτού του περίπλοκου προβλήματος και να βρούμε μία λύση έτσι ώστε τελικά να υπάρξει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα για την ψηφιακή οικονομία που είναι η πραγματική σημερινή οικονομία που θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε την πολυδιάσπαση των αγορών και θα μας επιτρέψει να ωφεληθούν οι συμμετέχοντες στις αγορές κάτω από δίκαιες και ισορροπημένες συνθήκες. Υπάρχουν δεδομένη πρόθεση των εισηγητών για να συνεργαστούν όλοι έτσι ώστε να βρεθεί μια ικανοποιητική λύση. Ευχαριστώ πολύ, Γκαμπριέλ. Ο κύριος Σύρφωξ εκ μέρους του ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έρχονται σε κατάλληλη στιγμή αυτές οι προτάσεις και πρέπει η Επιτροπή μα να τις εξετάσει προσεκτικά. Είμαστε σε μια εποχή που αυξάνεται η ψηφιακή παρουσία και το θέμα της φορολόγησης γίνεται φιλοσοφικό θέμα. Ε, εφόσον ε, οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε κράτη-μέλη χωρίς να έχουν φυσική παρουσία. Πιστεύω ότι πρέπει η έκθεση μας ε, να ορίσει τα κριτήρια για το τι σημαίνει σημαντική ψηφιακή παρουσία. Ιδανικά, χρειαζόμαστε μια διεθνή λύση στο πλαίσιο μιας ε, διεθνούς συμφωνίας για τη μεταρρύθμιση της φορολογίας εταιριών. Αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνο και καταλαβαίνω το σκεπτικό της Επιτροπής να διασφαλίσει ένα πεδίο θεμητού ανταγωνισμού το συντομότερο δυνατόν. Όσον αφορά τις επιπτώσεις τώρα στη φορολογία μεταξύ ε, εταιριών με φυσική παρουσία και εταιριών ε, με ψηφιακή παρουσία, θα ήθελα να φροντίσουν οι εισηγητές να εξασφαλίσουν την αναλογικότητα και να μην πέσουμε σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης κατά των μικρών ψηφιακών επιχειρήσεων. Το μήνυμά μας πρέπει να είναι ότι καλωσορίζουμε τις ε, εταιρείε που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στις χώρες μας. θέλουμε να συνεργαστούμε με, τους, με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές ώστε να υπάρξει και εποπτεία στα κράτη-μέλη και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζουμε αυτή την πρόταση της Επιτροπής ε, που την περιμέναμε εξάλλου εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. προσπαθεί να μπει σε μία ε, συζήτηση για τη φορολογία που έχει ξεκινήσει από τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά δεν πρόκειται καθόλου περί αυτού. Ε, δυστυχώς έχει καθυστερήσει αυτή η πρόταση. Θα πρέπει να την είχαμε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και βλέπουμε τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν με τη φορολογία των ψηφιακών εταιριών. ανοίγει πολύ, ε, όλο και περισσότερο η ψαλίδα μεταξύ των παραδοσιακών εταιριών και των εταιριών με ψηφιακή παρουσία. Η πρόταση της Επιτροπής ε, προσπαθεί να αντιμετωπίσει ε, αυτό το χάσμα μεταξύ των δύο τύπων εταιριών, φορολογώντας τις εταιρείες εκεί όπου δημιουργείται η αξία. Η ομάδα του Επιτρόπου Μοσκοβισή έχει συγκεντρώσει στοιχεία που δείχνουν ότι οι ψηφιακές εταιρείες πληρώνουν 9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με τις άλλες εταιρείες που πληρώνουν 23% φόρο. Το Facebook είχε φορολογικό συντελεστή 5% σε χώρες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, αν και πάνω από 50% των εσόδων του προέρχονται από υπηρεσίες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι δίκαιη λοιπόν αυτή η κατάσταση και διαταράσσει την εσωτερική αγορά. Κατανοώ βέβαια κάποιες ανησυχίες ότι η πρόταση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει φραγμό στην καινοτομία. Νομίζω ότι η σωστή νομοθεσία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της καινοτομίας. Θέλουμε ε, να έχουμε μια σωστή πρόταση αποφεύγοντας την γραφειοκρατία. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι όπως πάντοτε να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ, σε αυτή την περίπτωση, μεταξύ της δίκαιης φορολογίας και της ενθάρρυνσης της καινοτομίας. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεχτεί την πρόκληση αυτή. Το όριο ή τα όρια που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βοηθήσουν ε, τις νεοφυείς επιχειρήσεις ε, να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους χωρίς να τους επιβάλλουν υπερβολικές επιβαρύνσεις ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ε, στην έννοια του εντοπισμού του χρήστη που αποτελεί έννοια κεντρικής σημασίας για αυτό το νομοθετικό κείμενο. Εδώ υπάρχουν θέματα και τεχνικά και θέματα απορρίτου. Η φορολόγηση με βάση το γεωγραφικό σημείο στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης ε, βασίζεται στον εντοπισμό του χρήστη, το οποίο σημαίνει τήρηση στοιχείων για τους χρήστες και για την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται και τήρηση, διατήρηση αυτών των στοιχείων. Αυτό θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις του κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε με την Επιτροπή. Κλείνοντας, Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τη θέση μου ότι αν έχουμε δίκαιη φορολογία για την ψηφιακή παρουσία, θα είναι σημαντικό στοιχείο για να διευρύνουμε τα ωφέλη της παγκοσμιοποίησης και να ε, μειώσουμε το δυνατόν τη σκοτεινή πλευρά της παγκοσμιοποίησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Πίτερ. Δεν βλέπω κάποιον από τους πράσινους να ζητά να παρέμβει. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον σκιώδη της Γκουε, τον κύριο Σέρτοβαν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, τις παρεμβάσεις και τα ενδιαφέροντα ερωτήματα που τέθηκαν. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε λίγο πριν από το καλοκαίρι εκτιμά ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 20% των φορολογικών εσόδων χάνονται από τις ψηφιακές εταιρείες και είναι πάρα πολύ σημαντικό το, πάρα πολύ σημαντικό το μερίδιο αυτής της απώλειας το οποίο επομίζονται η Facebook, η Amazon, η Apple. Γι' αυτό και στο G20 από το 2015 συζητείται το θέμα αυτό ε, όσον αφορά ε, το θέμα, τις συζητήσεις που γίνονται γύρω από το BEPS, αυτήν την μεταφορά ε, εντός του ιδίου ομίλου κερδών από τη μία χώρα στην άλλη. Αντίστοιχες ε, συζητήσεις ε, υπάρχουν και στις ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια, γι' αυτό και ως αριστερά καλωσορίζουμε το γεγονός ότι πλέον έχει ξεκινήσει η σχετική συζήτηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε είπαν και προηγούμενοι ομιλητές ότι οι μεγάλες εταιρείες οι μεγάλες χώρες μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ενδιαφέρονται να καταλήξουν ή δυνατόν ακόμη και ω το τέλος του έτους σε μια γενική συμφωνία. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες φωνές, ιδίως από τις μικρότερες χώρες. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουν οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις. Ε, καθώς ε, τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για ζητήματα φορολογίας. Παρ' όλα αυτά, με θάρρο εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι πρέπει να συμβάλλουμε στη συζήτηση αυτή με θετικέ προτάσει προκειμένου να ε, επιτύχουμε ε, τουλάχιστον ε, την μεγαλύτερη φορολογική δικαιοσύνη, την καταπολέμηση της φοροαποφυγής είναι άλλωστε κάτι το οποίο περιμένουν από μας οι πολίτες μας. Ταυτόχρονα όμως με αυτόν τον τρόπο μπορούμε επιτέλους να περάσουμε από τον 20ο στον 21ο αιώνα, ιδίως στο θέμα της φορολόγησης των εταιρεών και να πω και κάποιες ε, παρατηρήσεις που έχω, να θέσω και κάποια ερωτήματα ε, και να ασκήσω και κάποια κριτική, αλλά και ε, κάποιες θετικές παρατηρήσεις. Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό το ότι πλέον συστήνεται, προτείνεται μάλλον σύσταση υπηρεσίας η οποία θα ελέγχει και θα επιτηρεί αυτήν την ενδομιλική. Ε, μεταφορά κερδών. Βεβαίως πρέπει να εξασφαλιστεί η αποφυγή διπλής φορολόγηση. Ταυτόχρονα θετικά βλέπουμε την ε, ε, υποχρεωτική υποβολή φορολογικών δηλώσεων από τις μεγάλες εταιρείες. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια στοιχεία που μας ανησυχούν στην πρόταση. Πρώτον, θεωρούμε ότι ο στόχος που έχει τεθεί για την ε, ε, συλλογή 5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε φορολογικά έσοδα είναι μικρός αν λάβει κανείς υπόψη του το πόσα χρήματα έχουν διαρρεύσει και δεν έχουν συλλεγεί από τις φορολογικές αρχές τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι ε, αν τεθεί ε, ο όρος του, το κριτήριο του, κύκλου εργασιών αυτό θα είναι άδικο για κάποιες εταιρείες. Το 3% για την Google για παράδειγμα είναι πάρα πολύ χαμηλό. Ενώ για άλλες εταιρείες, μπορεί, ιδίως τις μικρότερες, μπορεί να είναι πάρα πολύ υψηλό. Ε, Όμω είπε και ο εισηγητή ότι όλα αυτά τα θέματα είναι ανοιχτά, μπορούμε να τα συζητήσουμε και εμεί με τέτοιο ανοιχτό πνεύμα θα προσέλθουμε στη συζήτηση. Σε τελική ανάλυση θεωρούμε όμω ότι η αποτελεσματικότητα τη φορολόγηση, έτσι όπω προτείνεται, δεν είναι ε, ιδιαίτερα υψηλή. Όσον αφορά τις ε, συμπεριφορές μονοπολι... τις ή ολιγοπωλιακέ ορισμένων εταιρεών, ε, πρέπει κανείς να θεωρήσει δεδομένο ότι ενδεχομένως θα υπάρξει μετακύληση των επιπλέον αυτών φορολογικών εσόδων που θα θεσπιστούν σε άλλους, σε, άλλους, σε προμηθευτές, σε άλλες εταιρείες ή και στον τελικό ε, χρήστη. Και επίσης ε, δεν βλέπουμε τους, τους λόγους με τους οποίους αντιληγούνται ε, δεν συμφωνούμε με του λόγου με του οποίου αιτιολογούνται ορισμένε εξαιρέσει, όπω για το Spotify για παράδειγμα. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι πρέπει να θεσπιστεί τουλάχιστον μια ελάχιστη ε, φορολόγηση όλων των ε, εταιριών. Κάτι που άλλωστε είναι δεδομένο και ε, πρακτική και για άλλε άλλες που δραστηριοποιούνται σε άλλους κλάδου. Ο κύριος Βάλλη για το EFDD και εγώ να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον τους εισηγητές για τις παρεμβάσεις τους. Τα τελευταία χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει το θέμα επανειλημμένα και για την πολιτική είναι μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις η φορολογία των μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο πολλές φορές από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Συνεπώς λοιπόν η φορολογική πολιτική στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από πλευράς μας. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να διεθνοποιήσουμε όσο μπορούμε την υπόθεση αυτή. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό και ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο διότι το ευρωπαϊκό επίπεδο αφ' αυτού είναι και αδιεθνές εκπροσωπώντας άνω των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών χρηστών. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε σε επίπεδο φορολογικό τις επαχειρήσεις αυτές τις ψηφιακές. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υποστηρίξιμες. Το βασικό πρόβλημα της Ευρώπης και της Ευρωζώνης είναι ότι ορισμένες ιδρυτικές χώρες όπως το Λουσεμβούργο και οι κάτω χώρες δεν ονοματίζονται σωστά, αλλά οι χώρες αυτές όπως και η Ιρλανδία αντιτίθενται σε προτάσεις που γίνονται. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναζητήσει μία λύση για να μπορέσει να πιέσει τις χώρες αυτές οι οποίες αντικειμενικά δημιουργούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και να προσπαθήσουμε να δούμε τι θα κάνουμε ιδιαίτερα σε επίπεδο χωρών οι οποίες είναι πιο συνεργάσιμες. Έχει φτάσει νομίζω η στιγμή να αγριέψουμε θα έλεγα γιατί διαφεύγουν οι επιχειρήσεις αυτές εκατοντάδες εκατομμύρια κατέτος ενώ οι πτωχοί πολίτες καλούνται να πληρώνουν φορολογία και ε, πολλές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το παίζουν δάσκαλοι είναι αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα. Δεν βλέπω κάποιον άλλον από το ENF, οπότε ξεκινάμε τη διαδικασία του Catch the Eye. Είναι σημαντικό το θέμα, κάποιοι θα ήθελαν ίσως να πάρουν μέρος στη συζήτηση. Έχω αρκετές ερωτήσεις σε σχέση με την υπόθεση αυτή που μπορεί να απαντήσει ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που συνδέονται με κάποιες από τις παρεμβάσεις. Όταν μιλάμε με το θέμα της, κατανο... της κατανομής των... της φορολογικής δραστηριότητας επί των κερδών, ε, σε ποιο βαθμό μπορεί να αυξήσει τη φορολογία εις βάρος ορισμένων επιχειρήσεων. Νομίζω ότι επίσης εδώ το θέμα της ε, αποφυγής της διπλής φορολογίας είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη. Ε, σε ποιο βαθμό υπάρχει κίνδυνος διπλής φορολογίας και αν έχει αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος αυτός. Το δεύτερο θέμα είναι αυτό το οποίο έθεσε ο Ντάριος. Μιλάμε για την ψηφιακή οικονομία, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Νομίζω ότι η δίκαιη κατανομή των ε, φόρων δεν είναι κάτι το οποίο ανήκει αποκλειστικά στην ψηφιακή δραστηριότητα. Νομίζω ότι υπάρχει γενικότερα το θέμα των πωλήσεων εξαποστάσεων. επί επίσης. Ε, δημιουργούνται εδώ, χωρίς φυσική παρουσία, δυνατότητες ε, πρόσκλησης κερδών ε, από επιχειρήσεις. Συνεπώς λοιπόν νομίζω ότι η εμβέλεια των προτάσεων αυτών θα πρέπει να είναι ευρύτερη και να καλύψει επίσης και τις πωλήσει εξ Και τέλος Προφανώς ο φόρος αυτός ε, επί του κύκλου των επιχειρήσεων είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει, να λειτουργήσει σαν πλαίσιο αναφοράς, αλλά μερικές φορές μπορεί να είναι είτε υψηλότερο είτε χαμηλότερο από τη σωστή φορολογία που θα πρέπει να επιβληθεί. Αν είμαστε σε θέση να κατανείμουμε σωστά ε, τα έσοδα από την ψηφία οικονομία και από την ε, από τις πωλήσει ε, εξ αποστάσεως, ε, τότε θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες ε, ρυθμίσεις έτσι ώστε να μην είμαστε αρκετοί. Δεν θέλω να με παρανοήσετε. Θεωρώ παρόλα αυτά ότι η πρόταση που γίνεται από πλευρά σας είναι καλή. Ε, ίσως έχει καθυστερήσει κιόλας. Δεν θα πρέπει να αγνοηθεί το μέγεθος του προβλήματος και νομίζω ότι αν συνεχιστούν οι καταστάσεις αυτές θα οδηγήσουν σε πολύ αρνητικές καταστάσεις, ακόμα περισσότερο αρνητικές. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος θέλει το λόγο και θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. να παρουσιάσει τις θέσεις της και να αντιδράσει σε κάποιες από τις παρατηρήσεις που έγιναν. Ευχαριστώ πολύ. Θα περιοριστώ σε κάποιες απαντήσεις που θέλω να δώσω στα ερωτήματα που άκουσα. Θα ξεκινήσω με τη σημαντική ψηφιακή παρουσία. Τέθηκε ένα ερώτημα όσον αφορά τους δείκτες, αυτά τα όρια και πώς ακριβώς καθορίστηκαν αυτά. Το σημαντικό που πρέπει κανείς να έχει υπόψη του σε σχέση με αυτή την πρόταση είναι ότι ενδεχομένως Βεβαίω, σήμερα κάποιες από αυτέ τι μεγάλε εταιρείε έχουν ε, παρουσία φυσική σε μία χώρα ε, ή και καθόλου. Αλλά η ψηφιακή παρουσία θα είναι διαφορετική ε, σε κάθε χώρα και αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να ανταποκριθούμε, να απαντήσουμε. Η φυσική παρουσία ε, σε μια ε, χώρα ε, κοστίζει περίπου 60 με 80 χιλιάδες τουλάχιστον ευρώ το χρόνο. Θέλαμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι οι, οι εταιρείε θα έχουν και τη δυνατότητα να πληρώσουν αυτό το, αυτή τη φυσική τους παρουσία. Γι' αυτό και ορίσαμε αυτό το 3%. Να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι μια, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε ένα συγκεκριμένο χώρο ε, θα μπορεί να έχει και μια επαρκή ε, κερδοφορία. Γι' αυτό και θέσαμε ένα σχετικά ε, και θεωρούμε επαρκώς υψηλό όριο. Για τον φόρο επί των ψηφιακών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το τελευταίο ερώτημα που, ακούστηκε. Γιατί επιλέξαμε φόρο επί ε, του, κύκλου, εργασιών. Σημαντικό είναι να έχει κανείς υπόψη του ότι κατά τον σχεδιασμό αυτού του φόρου αντιμετωπίζουμε πάρα πολλούς περιορισμούς. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας βεβαίως το διεθνές ε, νομικό πλαίσιο Πρέπει να, ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις θεμελιώδεις ε, ε, ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους κανόνες του ΠΟΕ και εξαιτίας όλων αυτών των περιορισμών δεν είχαμε, πρέπει να σας πω, πάρα πολλές επιλογές στη διάθεσή μας. Ο φόρος κύκλου εργασιών, λοιπόν, ήταν κάτι που επελέγει ως εφικτή δυνατότητα. Βεβαίως προτιμούμε την φορολόγηση των κερδών, αλλά με τις ε, ψηφιακές εταιρείες, ε, αλλά και με τον, ε, φόρο επί των κερδών, στην ουσία ε, βρίσκεσαι διαρκώς στο ίδιο σημείο χωρίς να μπορείς να προχωρήσεις. Γι' αυτό και δεν επιλέγει ως μεταβατική λύση η συγκεκριμένη. Θέλαμε επίσης ο φόρος αυτός να είναι απλός, εύκολα εφαρμόσιμος, γιατί από τη φύση του πρόκειται για, μια μεταβατική, ε, για ένα μεταβατικό ε, μέτρο, γι' αυτό και δεν επιλέξαμε διαφοροποιημένα ε, φορολογικά επίπεδα. Θέλαμε να εξασφαλίσουμε ίσους όρους για όλες τις χώρες και ακριβώς επειδή δεν λάβαμε υπόψη μας το κόστος που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι εταιρείε, θεωρήσαμε ότι το 3% είναι μια ισορροπημένη λύση. Δεν είναι υπερβολικά υψηλό. Ε, δεν θέλαμε, ε, για παράδειγμα, να αποκλείσουμε ε, χώρες, ε, εταιρείες χαμηλής κερδοφορίας ή ακόμη και ζημιογόνες αν και συνήθως η συζήτηση επικεντρώνεται στις εξόχως κερδοφόρες εταιρείε. Γι' αυτό για να εξασφαλίσουμε αυτή την ισορροπία επιλέξαμε αυτό το όριο του 3%. Έπειτα. Κατανομή των κερδών και διαρθρωτικές λύσεις. και γιατί ε, βασίσαμε την πρότασή μας στους παλιούς κανόνες. Στόχος μας ήταν να, προσαρμόσουμε τους παλιούς κανόνες αυτό που, ε, αυτά που ισχύουν ε, για την μεταβίβαση των τιμών και αυτό είναι διαφορετικό σε σχέση με το CCTB. Στο CCTB καταργούνται όλα αυτά, διευκολύνεται η συμμόρφωση για τις εταιρείε, αλλά βεβαίως και μειώνεται η δυνατότητα να ε, μεταφέρει τα κέρδη σου σε χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Η CCCTB, ωστόσο, δεν αφορά όλε τι εταιρείε, αφορά μόνο τι εταιρείε με κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ κατ' έτος και γι' αυτό και θέλαμε να προτείνουμε κάτι που θα εμπεριέχει και τι άλλε εταιρείε που δεν περιέχονται στο CCCTB. Άλλωστε τέτοια εντολή είχαμε και από το Συμβούλιο για να υποβάλουμε μια πρόταση η οποία θα κινείται στο πλαίσιο του Διεθνού φορολογικού ε, συστήματος. κατά κάποιο τρόπο λοιπόν η πρότασή μα διατηρεί ε, την, ε, τους ισχύοντες κανόνες όσον αφορά τη λειτουργική ανάλυση και την αποφυγή μεταφοράς κερδών από τη μία χώρα στην άλλη. Θελήσαμε όμως να επικαιροποιήσουμε ε, τους κανόνες αυτούς λαμβάνοντας υπόψη και τη συμβολή των χρηστών στην παραγωγή αξίας. Έπειτα, τέθηκε ένα ερώτημα σε σχέση με τη μετακύληση των νέων, του νέου κόστους που θα δημιουργηθεί από τη φορολόγηση σε άλλες εταιρείες ή στους τελικούς χρήστες. Η απάντησή μας είναι απλή. Ναι, κάτι τέτοιο είναι πιθανό να συμβεί. Όπως άλλωστε κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και με κάθε άλλο φόρο που θεσπίζεται. Δεν μας ανησυχεί όμως. Η ανησυχία μας είναι οι εταιρείε μας να πληρώνουν τους ίδιους φόρους με τους, με τους υπόλοιπους. Να υπάρχουν ίσοι όροι σε αυτό το θέμα. Τώρα, αν μετακυλιστούν φορολογικά βάρη στους ε, τελικούς χρήστες ή σε εταιρείε που συνεργάζονται με αυτέ τι ε, μεγάλες ψηφιακέ εταιρείε, είναι κάτι που, που, μπορεί πράγματι να συμβεί. Αλλά δεν μας ε, ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει και κύριο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ίσου όρου ανταγωνισμού και δίκαιο σύστημα όσον αφορά τις εταιρείε μας. Αυτά να δώσω το λόγο τώρα στον συνάδελφο μου τον Μπάρτ για να μας μιλήσει λίγο για τον ορισμό των ψηφιακών υπηρεσιών και τον ορισμό της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας. Ευχαριστώ πολύ. Σημαντική ψηφιακή παρουσία. Τι συνιστά σημαντική ψηφιακή παρουσία. Πρώτον, θα πρέπει να υπάρχει ε, διαδικτυακή διεπαφή, δηλαδή ιστοσελίδα ή εφαρμογή που πρέπει να είναι προσβάσιμη στους χρήστες και από εκεί να παρέχονται ψηφιακές υπηρεσίες. Για τον ορισμό των ψηφιακών υπηρεσιών βασιστήκαμε ή μάλλον αντιγράψαμε τον ορισμό από τον κανονισμό για το ΦΠΑ του 2011, συγκεκριμένα το άρθρο 7. Ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, δηλαδή υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου, που εξαρτώνται από την τεχνολογία με, που δεν απαιτούν παρά μόνο ελάχιστη παρέμβαση από τον χρήστη και από τον προμηθευτή και υπάρχει και ένας ολόκληρος κατάλογος όπου εξηγείται με λεπτομέρεια ποιες υπηρεσίες θεωρούνται ψηφιακές και ποιες υπηρεσίες δεν θεωρούνται ψηφιακές. Τα ψηφιοποιημένα προϊόντα βασικά εννοούμε ε, software, ε, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων ή ε, πρόσβαση σε εμπορικές αποθήκες. Αυτά είναι ψηφιακές υπηρεσίες. Όχι όταν κάποιο προϊόν, υλικό αγαθό παρέχεται απλά μέσω διαδικτυακής παραγγελίας. Βασιστήκαμε λοιπόν σε έννοιες που έχουν καθιερωθεί, που έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο εδώ και χρόνια και που είναι γνωστές και στις φορολογικές αρχές και στους φορολογούμενους πολίτες. Για την κατανομή των ε, κερδών και τη CCTB. Θεωρούμε ότι η CCTB θα πρέπει να συμπεριλάβει και εκείνη την έννοια της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας μια είναι η οποία θα πρέπει και να αναπροσαρμόζεται για να λαμβάνονται υπόψη και οι εξελίξεις όσον αφορά τις ψηφιακές εταιρείες. Επιτρέψτε μου ε, να επανέλθω, γιατί νομίζω ξέχασα να απαντήσω. Ρωτήσατε αν πρόκειται για ζήτημα κατανομής ε, της φορολόγησης ή ζήτημα αύξησης της φορολόγησης. Η απάντηση είναι ότι είναι λίγο και από τα δύο. Η πρόταση για τη σημαντική ψηφιακή παρουσία θα ανακατανείμει τους φόρους με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή θα υπάρξει μια διαφορά όσον αφορά το πού θα πληρώνουν οι εταιρείε τους φόρους τους, αλλά θα υπάρξει και μια αύξηση των φόρων που θα πληρώνουν. Γιατί δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα τεχνητά να μεταφέρονται κέρδη σε ε, δικαιοδοσίες φορολογικές με χαμηλότερους συντελεστές. Ε, ε, ρωτήσατε επίσης ε, θέσατε το θέμα ότι η δίκη φορολόγηση δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την ψηφιακή οικονομία. Έχετε δίκιο και εδώ σας παραπέμπω στην πρότασή μας για την CCCTB που θεωρούμε ότι απαντά σε αυτό το θέμα ε, ιδίως όσον αφορά τις εξαποστάσεις, εξαποστάσεως πωλήσει. και αν κανείς ε, ε, συνυπολογίσει και συνεκτιμήσει και τη CCTV και την πρόταση για τη σημαντική ψηφιακή παρουσία νομίζω ότι δίνεται μια καλή απάντηση διότι ε, ένας από τους ε, παράγοντες που λαμβάνονται επόψη στην εξίσωση και στον μαθηματικό τύπο αυτό είναι και η, φυσική απόσταση σε μια εξαποστάσεως πώληση. Uh, Και τώρα να δώσω το λόγο στους συζητητές, αν θέλετε, για λίγα λεπτά. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν στην ε, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Έχω τρία-τέσσερα σημεία τα οποία θα αναφέρω πολύ σύντομα. ο σκοπός μας ε, είναι να εξασφαλίσουμε δίκαιο πεδίο ανταγωνισμού για όλους και να έχουμε μεγαλύτερη δικαιοσύνη στο φορολογικό σύστημα. Όσοι είναι κατά της πρωτοβουλίας αυτής θα πρέπει να σταθμίσουν ε, τα επιχειρήματα αυτά, διότι αν δεν κάνουμε τίποτα θα είναι σαν να συμφωνούμε με το τωρινό σύστημα, το οποίο όπως πολλοί προηγούμενοι ομιλητές είπαν, δεν είναι κατά κανένα τρόπο τέλειο. Δεν διασφαλίζει την δικαιοσύνη και αφήνει πολλές δυνατότητες αποφυγής φορολογίας, ιδιαίτερα για τους μεγάλους φορολογουμένους. Αυτό να το έχουμε κατά νου, γιατί αν συμφωνήσουμε επί αυτής της γενικής αρχής, τις λεπτομέρειες νομίζω μπορούμε να τις βρούμε. Αλλά υπενθυμίζω ότι ο στόχος μας είναι στο τέλος της διαδικασίας αυτής να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα που θα εξασφαλίζει ένα δίκαιο πεδίο ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείε. Δεύτερον, η πρότασή μας αυτή δεν θέλει να φορολογήσει οτιδήποτε ψηφιακό υπάρχει, γιατί η οικονομία μας, η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, είναι ψηφιακή στο σύνολό της. Και υπάρχουν πολλοί φόροι, ε, πολλές δραστηριότητες που δεν ε, ε, φορολογούνται με βάση αυτή την πρόταση. Οι πωλήσει μέσω διαδικτύου, παραδείγματο χάρη, δεν φορολογούνται από τον νέο αυτό μέσο το οποίο προτείνουμε. Ο στόχος της Επιτροπής, όπως εγώ τον αντιλαμβάνομαι, είναι η παροχή υπηρεσιών που δεν θα είχαν φορολογηθεί καθόλου αν δεν βάζαμε αυτό το φόρο στις ψηφιακές υπηρεσίες. Τώρα όσον αφορά την κατανομή του φόρου έναντι αυξήσεων φόρου, έδωσε μια απάντηση εκπρόσωπος της Επιτροπής και συμφωνώ. Θέλουμε να έχουμε δίκαιη κατανομή των φορολογικών υποχρεώσεων και σε κάποιες δραστηριότητες έχουμε αύξηση του φόρου. Για κάποιες δραστηριότητες για πρώτη φορά ε, επιβάλλεται φορολογία και για κάποιες άλλες αυξάνεται ο φόρος διότι δεν θα έχουν πλέον οι εταιρείε τη δυνατότητα να μεταφέρουν ε, την ε, φορολογική τους υποχρέωση σε δικαιοδοσίες με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Όπως και με όλους τους έμεσους φόρους ε, ε, για να αντιμετωπίσουμε την ε, άδικη φορολόγηση. Ε, θέλουμε να επιβάλλουμε δίκαια μέτρα για να μην επιβαρύνονται οι καταναλωτές. Αν βελτιώνουμε τον ανταγωνισμό, θα προσπαθήσουν οι εταιρείε να αυξάνουν το μερίδιο της αγοράς τους και δεν θα υπάρχουν αθέμητες πρακτικές και επιβάρυνση των φορολογουμένων. Η φορολογία πάντοτε έχει ένα θετικό αποτέλεσμα διότι φέρνει έσοδο στον προπολογισμό και ένα αρνητικό διότι μειώνει το εύρος των δραστηριοτήτων που θα ήταν ε, ευρύτερες αν δεν φορολογούνταν. Αλλά πρέπει να βρούμε πάντοτε την κατάλληλη ισορροπία. Ευχαριστώ πολύ. Πολ, θέλεις το λόγο? Ναι, θα είμαι κι εγώ σύντομο. Συμφωνώ με τον Τάριο Ροζάτη ότι αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε αποτελεσματική και δίκαιη φορολόγηση. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Ακούγοντας τη συζήτηση, νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι εδώ αντιμετωπίζουμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Και πριν από τις εκλογές πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. Εταιρείε όπως η Google και η Facebook που έχουν ε, μεγάλα κέρδη, είναι από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, δεν μπορεί να μην πληρώνουν φόρους. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Άκουσα και κάποια θέματα που αφορούν την υλοποίηση και όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας γιατί βρισκόμαστε σε ε, νέο έδαφος, ε, χαρτογράφητο έδαφος και θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε με βάση αυτό που έχει προτείνει η Επιτροπή για, την για τον ψηφιακό τομέα, ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και γενικότερα για τον φόρο εταιριών, ώστε να καταλήξουμε σε μία εφικτή ε, λύση η οποία θα μας δώσει αποτελέσματα σε αυτό το νέο τομέα στον οποίο κινούμεθα. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της αδικίας και της μη αποτελεσματικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, ε, Ευχαριστώ τους εισηγητές ε, και την Επιτροπή και όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Ε, να σας πω για το χρονοδιάγραμμα ότι θα έχουμε μια δημόσια ακρόαση τον Σεπτέμβριο, θα 10 Σεπτεμβρίου, θα εξεταστεί το σχέδιο έκθεση στις 9 Οκτωβρίου, υποβολή τροπολογιών μέχρι 16 Οκτωβρίου, που θα εξεταστούν μέχρι 19 Νοεμβρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 3 Δεκεμβρίου και στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τα σημεία 7 και 8 και περνάμε τώρα κατευθείαν σε, στα δύο επόμενα σημεία για τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις. Δύο εκθέσεις, Ashley Fox από τη ΣΙΑΡ και η Καρολίν Νάκτεγκαλ από τους Φιλελευθέρους. Και έχουμε και πολλούς σκιώδη εισηγητές. Γι' αυτό η γραμματεία έχει προτείνει μέχρι 8 λεπτά για κάθε εισηγητή και δίνω το λόγο στον Ashley Φόξ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση κανονισμού για την πλήθο χρηματοδότηση για το crowdfunding είναι πολύ σημαντική. Μετά την κρίση, η Επιτροπή μας έχει προτείνει ε, νομοθεσία κυρίως για να αυξηθεί η ρύθμιση ε, σχετικά με τις δανειοδοτήσεις προς επιχειρήσεις. Παράλληλα, έχουμε κάνει βήματα και για την ε, εναλλακτική χρηματοδότηση και για τη δημιουργία Ένωσης Κεφαλαίου Η παρούσα πρόταση αυτό θέλει να επιτύχει και γι' αυτό χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής. Υπάρχουν διαφορετικά καθεστώτα στην ενιαία αγορά, τα οποία παρεμποδίζουν τη διασυνοριακή δραστηριότητα και Γι' αυτό με, μια, ε, με ένα ευρωπαϊκό καθεστώς, μια ευρωπαϊκή πρόταση, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις διασυνοριακές δραστηριότητε στην Ευρώπη χωρίς να επηρεάζουμε τις ε, εθνικές διατάξεις. Καταλαβαίνω ότι χρειάζονται κάποιες αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής για να έχουμε το βέλτιστο όφελος. Στο σχέδιο έκθεση το οποίο έχω ετοιμάσει, νομίζω ότι υπάρχουν πέντε τομείς στους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχήν, το όριο για τις ε, προσφορές crowdfunding, η εποπτεία από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, η διαφοροποίηση μεταξύ απλής και πολύπλοκης δομής ε, πληθοχρηματοδότησης, ε, οι αρχικές προσφορές εικονικού νομίσματος και η δημιουργία πλατφόρμας που θα είναι δίκαιη και για φορείς από τρίτες χώρες για το όριο από 1 εκατομμύριο προτείνω να αυξηθεί στα 8 εκατομμύρια ώστε να ευθυγραμμιστεί με την οδηγία για το ενημερωτικό δελτίο. Και στις δύο οδηγίες θα θέλει να υπάρχουν παρόμοιες διατάξεις. Τα 8 εκατομμύρια πιστεύω για λόγους συνέπειας είναι σωστή επιλογή. Η αύξηση αυτού ορίου θα κάνει την πρόταση αυτή πιο ελκυστική διότι κάποια εθνικά καθεστώτα ήδη έχουν υψηλότερο όριο. Τώρα, όσον αφορά την εποπτεία και την αδειοδότηση των παρόχων υπηρεσιών crowdfunding, δεν νομίζω ότι θα πρέπει όλες αυτές οι πλατφόρμες να ε, επιβλέπονται μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει εμπειρία στις εθνικές αρχές και θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνεπής εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Επίσης, ε, η... ο τομέας αυτός των παρόχων υπηρεσιών crowdfunding μπορεί να είναι ε, ιδιαίτερα πολύπλοκος και θέλω να κάνουμε τη διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των πλατφορμών ε, που ε, έχουν που διευκολύνουν τη σύζευξη επενδυτών και κυρίων των έργων και των πλατφορμών που καθορίζουν την τιμολόγηση και την ομοδοποίηση προσφορών με καθορισμό διαφορετικών απαιτήσεων γνωστοποίησης για κάθε κατηγορία θέλω να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την πρόταση για να δημιουργηθεί ε, και κάποια ρύθμιση για τις αρχικές προσφορές εικονικού νομίσματος. Δεν έχουμε μια οριστική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Αναγνωρίζουμε την δουλειά που έχει γίνει από, τους, από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και από την ΕΣΜΑ και από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία και τουλάχιστον να προτείνουμε μια προσωρινή λύση. Το σχέδιο εκθεσής μου προτείνει ε, να ε, αφορά ε, αυτό το οποίο θα, θα προτείνουμε, τις αρχικές προσφορές εικονικού νομίσματος, αποκλείοντας αυτούς που δεν λειτουργούν με κάποιο ομόλογο ούτε, ώστε να έχουμε πρότυπα και μέτρα προστασίας σε σχέση με τις προσφορές αυτές που θα αποτελούν μια εξαιρετική ροή χρηματοδότησης για νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας. Πιστεύω ότι ε, αυτές οι πλατφόρμες που συζητάμε είναι εξαιρετική ευκαιρία για να ε, ε, επεκταθούμε πέραν της ενιαίας αγοράς. Αυτό θα είναι ευκαιρία επενδύσεων για αυτά τα έργα και θα διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι επενδυτές έχουν την ίδια προστασία όταν επενδύουν σε τρίτες χώρες. Αυτό θα ε, καταστεί δυνατό με αδειοδότηση προς τρίτες χώρες για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα διαβατήριο, ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο για την ευρωπαϊκή αγορά. Είμαστε πολύ φιλόδοξοι για το χρονοδιάγραμμά μα. Θέλουμε την έκθεση να τη συζητήσουμε στην Επιτροπή τον Νοέμβριο και προσβλέπω στη συνεργασία με την συνεισηγήτρια και τους σκιώδεις συζητητέ. Είδατε ότι ήμουν σύντομο, μόνο πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Άσλη, και ευχαριστούμε ε, που ε, θα συζητηθεί αυτή η έκθεση στο συντομότερο δυνατόν και δίνουμε το λόγο ε, στην Ναθγκαλ από το ΑΛΔΕ. Για μένα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, αντιμετωπίζουν την δυνατότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας, ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων απασχολείται στις μικρομεσαίες. Γνωρίζουμε όμως ότι καμία πόλη και κανένα χωριό δεν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τις μικρομεσαίες. Υπάρχει βέβαια οι μεγάλες επιχειρήσεις αλλά οι μικρομεσαίες σε τοπικό επίπεδο παίζουν καθοριστικό ρόλο, αντιπροσωπεύουν θα έλεγα την επιχειρηματικότητα της κοινωνίας μας και πολλές φορές δημιουργούν θέσεις εργασίας καθημερινά. Ε, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες φιλόδοξοι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν συνεχώς δυσκολίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν οφείλει να τους βοηθήσει. Οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, δεν περιορίζονται μόνο σε τοπικό γεωγραφικά επίπεδο και ο ρόλος τους θα πρέπει να διευκρινιστεί καλύτερα. Και εδώ τίθεται το θέμα του crowdfunding. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τις νεοπαγές, νεοπαγείς αυτές επιχειρήσεις ε, πέραν του παραδοσιακού ε, τύπου ε, δανειοδότησης που πολλές φορές τοπικά δεν λειτουργεί. Θα πρέπει να υπάρξουν λοιπόν πρέπει να υπάρξει στήριξη των προσπαθειών crowdfunding και των διασυνοριακών μορφών crowdfunding. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις για τις δυσκολίες αυτές μια επιχείρηση μπορεί να έχει μια καταπληκτική ιδέα για ένα νέο προϊόν και πρέπει να βοηθηθεί η επιχείρηση αυτή έτσι ώστε να συλλέξει ε, χρήματα από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό είναι θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι θετικό για τα κράτη-μέλη και τους πολίτες. Η πρόταση Fox λοιπόν είναι μια καλή πρόταση, συμφωνώ με τις περισσότερες προτάσεις του εισηγητή. Ε, οι προτάσεις οι οποίες γίνονται θα έλεγα είναι πάρα πολύ καλές. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να διευκολύνουμε επίσης ε, την χρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων. Είναι περίπλοκη η κατάσταση η οποία ισχύει σήμερα. Η έκθεσή μου για την οδηγία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Εγώ συμφωνώ με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χαιρετίζω τις επιμέρους προτάσεις. Θα συνεχίσουμε λοιπόν ε, την εξέταση των πραγμάτων αυτών στο μέλλον με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Ας περάσουμε τώρα στους σκιώδεις εισηγητές. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους εισηγητές για τις προτάσεις τις οποίες μας έχουν αποστείλει. Και εγώ είμαι ικανοποιημένη που θα αντιμετωπίσουμε το θέμα του crowdfunding που είναι ένας καινοτόμος ψηφιακός και προσβάσιμος τρόπος για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που καλούνται να παίξουν έναν βασικό ρόλο στο κοινοτικό έδαφος και που αντιπροσωπεύουν το 90% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να βοηθήσουμε να την χάνουν και περαιτέρω στήριξης. Αν θέλουμε να πετύχει η προσπάθεια αυτή, θα πρέπει, θα έλεγα, να διέπεται από κάποιες συγκεκριμένε αρχές. Αν θέλουμε να αναπτυχθεί το crowdfunding σε διασυνοριακό επίπεδο, θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα πλαίσιο, ε, να δημιουργήσουμε, συγγνώμη, ένα πλαίσιο κυρίως αποτελεσματικό και απλό. Συνεπώς λοιπόν το crowdfunding θα μπορέσει να προστατεύσει σωστά τους επενδυτές. Στην έκθεσή του ο κύριος Φόξ κάνει αρκετές προτάσεις. Κάποιες από τις προτάσεις αυτές φαίνονται πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όπως η αύξηση του ανωτάτου ορίου από 1 σε 8 εκατομμύρια ε, επίσης οι ιδέες τις οποίες καταθέτει ε, για το θέματα του μάρκετινγκ. Μια άλλη πρόταση επίσης, ε, την οποία έχει ήδη αναφέρει ο κύριος Φόξ και η οποία είναι σημαντική, περιλαμβάνει τις λεγόμενες αρχικές εκδόσεις c'est vrai qu'il n'y a pas encore de, de, de, de texte. De... Εικονικών νομισμάτων. Ε, νομίζω ότι εδώ σε αυτό τον τομέα είναι πάρα πολύ νωρίς να προχωρήσουμε με συγκεκριμένες λύσεις και έχω την αίσθηση ότι το κείμενο εδώ δεν είναι ε, το σωστό μέσο και ο σωστός χώρος. Έχω ε, εντοπίσει και κάποια άλλα επιμέρους θέματα τα οποία θα σας μεταφέρω σε σχέση με την επικοινωνία και το μάρκετινγκ και έχω επίσης ε, τονίσει ότι δεν θα πρέπει να έχουμε πολύ δύσκολους κανόνες έτσι ώστε να μην δυσκολεύουμε τα προγράμματα τα οποία προτείνουν οι πλατφόρμες αυτές. Υπάρχει και το θέμα της οικονομικής συμμετοχής ε, των εταιριών αυτών στα προγράμματα έχει σημασία αυτό γιατί είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τους επενδυτές και τους θεσμικούς μάλιστα επενδυτές. Να αναφερθώ επίσης και στην ανάγκη η οποία υπάρχει προσαρμογής ορισμένων διατάξεων σχετικά με το είδος των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων και των επενδυτικών δραστηριοτήτων. Εδώ υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες και θα πρέπει να γίνει η διάκριση. Τώρα, αν θέλουμε το crowdfunding να αναπτυχθεί στην Ευρώπη χωρίς εμπόδια, προβλήματα και σκάνδαλα, έχει σημασία αυτοί που επιλέγουν να επενδύσουν μέσω του crowdfunding να είναι σωστά ενημερωμένοι για τους κινδύνους τους οποίους ε, διατρέχουν ε, και για το ότι μπορεί να χάσουν τα χρήματά τους. Επίσης ε, τίθεται το θέμα του να προβλεφθούν εδώ κάποιες ρυθμίσεις για τις ισοτιμίες. Σε αυτή τη φάση των συζητήσεων δεν το βρίσκω απαραίτητο. Πάντως οι συζητήσεις οι οποίες έγιναν και θα συνεχιστούν είναι πλούσιες και επικοδομητικές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βαντεκέλα, δεύτερος σύντης. Ευχαριστώ πολύ. Ακούστηκαν ήδη πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια καταπληκτική ιδέα και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν την νεοπαγή εταιρεία που θέλουν να ιδρύσουν και ή δυνατόν να την εξελίξουν και σε ε, μεγαλύτερης κλίμακας εταιρεία. Αυτή η δυνατότητα πρέπει να υπάρχει και εδώ μπορεί να απαντήσει πραγματικά αυτή η διαδικασία της ε, συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ιδίως αυτό αφορά νέους ανθρώπους προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με αυτά που είπε η κυρία Σάντερ. Πρέπει αυτή η δυνατότητα να υπάρχει, να είναι απλή, να είναι εύκολη και πρέπει να υπάρχει και επαρκής προστασία των επενδυτών. Όσον αφορά την έκθεση της κυρίας Νάχταγκαλ, συμφωνώ ότι πρόκειται περί μιας ε, ευσύνοπτης ε, έκθεσης και εγώ υποστηρίζω αυτή την ε, προτροπή να υποστηριχθεί ε, η πρόταση της Κομισιόν. Αυτό θα κάνουμε και εμείς ως πολιτική ομάδα και ε, ελπίζουμε να καταλήξουμε σύντομα σε θέση του Κοινοβουλία. Και νομίζω ότι σε αυτό θα συμβάλλουμε όλοι οι σκιώδεις εισηγητές. Για τους σοσιαλιστές η κυρία Εύα Καηλή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να, συγχωρώ τον, να συγχαρώ τον Ashley Fox ε, και την κυρία Νάχτιγκαλ για το έργο τους. Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση, εξετάζουμε αυτόν, τον, ε, αυτή την πρόταση και τη δυνατότητα ε, μεταφοράς κεφαλαίων προς την πραγματική οικονομία προκειμένου να ενισχυθεί η ε, παραγωγικότητα συνολικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να ε, στεφθεί με επιτυχία αυτή η διαδικασία τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Καταρχά, χαιρετίζουμε την ε, πρόταση του εισηγητή να αυξηθεί το όριο από το 1 εκατομμύριο στα 8 εκατομμύρια για κάθε εκστρατεία πληθό χρηματοδότηση. Όσον αφορά το ACS ε, συμφωνούμε με την προσέγγιση που έχει υιοθετήσει ο εισηγητής, αν και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί σε μεγαλύτερο βάθο. Σε τεχνικό επίπεδο θα ήθελα να προσθέσω και κάποιες παρατηρήσεις. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, αυστηροί όσον αφορά την διαφάνεια, όσον αφορά την ε, προστασία των επενδυτών το, το επίπεδο ε, της χρηματοδότησης και πρέπει να υπάρξει προστασία από ασύμετρες ε, διαρροές ε, πληροφοριών ε, και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η προστασία των επενδυτών. Θα πρέπει να υπάρχουν διατάξεις οι, οποίοι, οι οποίες θα ε, υποχρεώνουν όλους, τους, ε, όλους εκείνους που δραστηριοποιούνται στην πληθροχρηματοδότηση να παρέχουν ε, με διαφάνεια τις πληροφορίες όποτε τους ζητούνται από τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά σε αυτό στον οικονομισμό. Η συμμετοχική χρηματοδότηση θα πρέπει να ε, εξασφαλίζει ε, την προστασία και των επενδυτών, των ανθρώπων που βάζουν τα χρήματά τους σε ε, τέτοιου είδους εκστρατείες και project και ε, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα πρέπει να, να, είναι εγγενές των ίδιων των, πλα, των πλατφορμών. Επίσης, η πληθυσματοδότηση δεν θα πρέπει να είναι επικίνδυνος, ε, επικίνδυνο μέσο χρηματοδότησης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Γι' αυτό και πρέπει να μειωθεί ε, και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος με τη θέσπιση συγκεκριμένων ασφαλιστικών δικλείδων και εχέγγυων γι' αυτόν. Και τέλος, θα πρέπει ε, οι πλατφόρμες αυτές να μην, να μην λειτουργούν ως δευτερογενής ε, σφαίρα χρηματοδότησης και να κάνουμε και μια πρόταση. Η πρόταση, η πρόταση της Κομισιόν ακολουθεί και τις προτάσεις που έχουμε βάλει εμείς ως Κοινοβούλιο. Ε, για μας ωστόσο ο ΕΣΜΑ πρέπει να ε, διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο ώστε να εξασφαλιστεί ότι το εναρμονισμένο περιβάλλον θα εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα της, ε, στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Πρέπει να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το ρόλο του ΕΣΜΑ και τέλος για, τα ισοδύναμα τρίτων, για τις ισοδύναμες ε, εταιρείε τρίτων χωρών χαιρετίζω την πρόταση, ωστόσο νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να συζητήσουμε για το πώς ακριβώς θα υλοποιηθούν αυτά στην πράξη. Αυτά προς το παρόν θα ήθελα να ξαναευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του και προσβλέπω στη συνεργασία μας και με τους ε, άλλους σκιώδεις εισηγητές και επειδή πρέπει να μιλήσω και για τον ε, δεύτερο φάκελο ένα πολύ σύντομο ε, σχόλιο δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα αν και θα θέλαμε να λάβουμε περισσότερες προφορίες όσον αφορά την οικονομική λογική που οδήγησε την Κομισιόν ε, ε, στο να αποκλείσει ε, τις εταιρείε που έχουν λάβει άδεια υπό την MIFID από τις διατάξεις της συγκεκριμένης πρότασης. Ευχαριστούμε πολύ Εύα. Ε, ο εισηγητής θέλει να, να μιλήσει. Βεβαίως να δώσω το λόγο πρώτα στους σκιώδεις αν υπάρχουν άλλοι. Πράσινοι δεν υπάρχει. Ε, ούτε από την ΚΟΕ, ο κύριος Βάλη από το EFTD. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για τις παρεμβάσεις τους, για τα όσα είπαν και για το έργο που ε, πρόκειται να επιτελέσουν. Όσον αφορά την πληθοχρηματοδότηση και τη σχετική πρόταση, θεωρούμε ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση γιατί θα ενισχύσει μια, ένα χρηματοδοτικό κανάλι που είναι πολύ σημαντικό για τις startup εταιρείε ε, για τις εταιρείε καινοτομία που πολλέ φορέ δεν έχουν πρόσβαση στην παραδοσιακή πίστοση και χρηματοδότηση. Όσον αφορά τα όρια που συζητήθηκαν και εδώ, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν τέτοια όρια, διότι όταν ε, κανείς προσπαθεί να βρει χρήματα και κεφάλαια από μη συμβατικού τρόπους, ε, θα πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένες ε, ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να, να, ανοιχνεύονται οι ροές των κεφαλαίων και να μην βρεθούμε σε καταστάσεις ε, ξεπλήματος βρώμικου χρήματος για παράδειγμα και γνωρίζουμε ότι αυτά τα καινοτόμα εργαλεία πολλές φορές χρησιμοποιούνται ε, και για τέτοιου είδους σκοπούς. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα ανείχνευσης και παρακολούθησης των ροών κεφαλαίων. Ε, θεωρώ όμως ότι τα όρια δεν είναι αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλιστεί κάτι τέτοιο, από μόνα τους τουλάχιστον. Όσον αφορά την επιτήρηση και την εποπτεία, θα προτιμούσαμε μια προσέγγιση που θα ενίσχυε το ρόλο των εθνικών αρχών παρά τη θέσπιση μιας, ε, ενός κεντρικού οργάνου. Ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν περισσότερη εμπειρογνωμονωσία, περισσότερες γνώσεις και πολύ αποτελεσματικότερα μπορούν να χειριστούν τα ζητήματα που θα ανακύπτουν και στο μέλλον. Όσον αφορά την επιλογή των έργων που χρηματοδοτούνται, κάποιες ε, Ιταλικές αρχές έχουν ήδη ε, αξιοποιήσει και εφαρμόσει κανόνες πληθοχρηματοδότησης. Κάτι που σημαίνει ότι εκείνοι που χρησιμοποιούν την συμμετοχική χρηματοδότηση το κάνουν ακριβώς γιατί δεν θέλουν να προσφύγουν στις τράπεζες για τη δανειοδότησή τους. Εκείνοι λοιπόν που θέλουν να συμμετέχουν και να ξεκινήσουν μια διαδικασία συμμετοχικής χρηματοδότησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι θα συμμετέχουν ε, και τράπεζες στη διαδικασία χρηματοδότησης αυτή τουλάχιστον έως το όριο του 5%. Εν πάση περιπτώσει αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. γεγονό πάντω είναι και σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε θέση του Κοινοβουλίου και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να καταλήξουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Κάτσε διά, κύριε Σαγκέρο. Um, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συζητητές για την ε, έκθεσή τους. Νομίζω ότι είναι καλές οι προτάσεις που συζητούμε και που ελπίζουμε να ενισχύσουν την ε, ε, ροή κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις νεοπαγείς εταιρείες. Έχουμε μια πρόταση η οποία θα είναι το 20, 29ο καθεστώς που θα αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι και στις δύο προτάσει θα υπάρχουν επαρκή κίνητρα και επαρκές επίπεδο προστασίας των επενδυτών. Και κάτι τελευταίο για τις ε, εταιρείες από τρίτες χώρες. Όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεδομένως ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και μια ε, ενιαία αγορά στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ε, θα προσελκύονται επενδυτές και από μέσα από την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και να δοθούν συγκεκριμένα κίνητρα προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστούμε Νένο. Δεν φαίνεται να ζητά κάποιος άλλος το λόγο. Επομένως θα δώσω το λόγο στους συζητητές. Καρολίνη Νακτεγκάλ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Προσβλέπω στη συνεργασία μαζί τους, συζητήσεις που θα έχουμε σχετικά με τις τρίτες χώρες. Θέλω πράγματι και εγώ να εμβαθύνουμε στη συζητήση μας στο θέμα αυτό. Είναι περίπλοκο. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια κοινά αποδεκτή λύση. Περιμένω λοιπόν να, γίνουν, να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις και ε, ελπίζω σύντομα να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη φάση. Ευχαριστώ ο κύριος Άσλι Φόξ, ο εισηγητής μας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και να ευχαριστήσω και την συνεισηγήτρια και τους σκιώδεις για τις παρεμβάσεις τους. Συμφωνώ με την Καρολάιν ε, και την ανάλυση της για την ανάγκη να δοθεί δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν ε, ε, να συγκεντρώνουν κεφάλαια ε, πιο εύκολα. Είναι ένα από τα ζητήματα που ανέκυψε μετά την, την κρίση και αυτή η πρόταση πραγματικά διευκολύνει μια τέτοια διαδικασία. Άννα Σάντερ, συμφωνώ μαζί σου ότι χρειαζόμαστε ένα απλό και ε, εύκολα εφαρμόσιμο σύστημα ξέρω ποιε είναι οι ανησυχίε που εξέφρασε όσον αφορά τη διατύπωση των προτάσεών, μας, των προτάσεών μου για τι ε, ICO. Και βεβαίω είμαι στη διάθεσή σου για να καταλήξουμε ενδεχομένω και σε κάποιε συμβαστικέ λύσει ε, για να βρούμε την καταλληλότερη διατύπωση. Εύα Καηλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ε, ενέταξες στα σχόλιά σου αυτούς τους ICO. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όλες τις πολιτικές ομάδες έθεσε το ζήτημα τη ε, διαφάνεια και τη προστασία των επενδυτών. Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι πολύ σημαντικά ζητήματα αυτά και θα περιμένω τι πολύ συγκεκριμένε προτάσει σου για να τις εντάξουμε στην έκθεσή μου. Κύριε ε, είπατε ότι θέλετε να υπερβείτε ε, το όριο των 8 εκατομμύριων. Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν ε, νομίζω ότι θα συγκέντρωνε πλειοψηφία. Α το συζητήσουμε όμω για να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Επίσης, ε, αναφερθήκατε στα ισοδύναμα τρίτων, τρίτων χωρών. Το θέμα αυτό καλύπτεται στην έκθεση, αλλά το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο τον Brexit το βασικό ζήτημα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η μικρομεσαία επιχείρηση μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τη, τη μεγαλύτερη δυνατότητα ε, χρηματοδότησης. Το αν ε, αυτό... αυτό, αυτό αφορά και τις ε, εταιρείε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις, ε, τις εταιρείες που ενδεχομένως έχουν την έδρα τους στην Ελβετία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Μάρτιο του 2019. Το ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει λοιπόν είναι πώς μπορεί να συγκεντρωθούν τα περισσότερα και τα μεγαλύτερα δυνατά κεφάλαια προκειμένου να κατευθυνθούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα το συζητήσουμε αυτό ε, όσον αφορά τη ρύθμιση των ICO. Και υπάρχει και σχετική διακομματική ε, ε, ομάδα που θα συνεδριάσει στις 4 Σεπτεμβρίου, στις 4.30 το απόγευμα, στην αίθουσα AP2. Ε, και με όλα αυτά ε, να σας πω ότι προσβλέπω και εγώ στην συνέχιση της επικοδομητικής μας συνεργασίας. Πρόεδρος, ωραία. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Λοιπόν, Όσοι θέλουν να συζητήσουν το θέμα αυτό σε μεγαλύτερο βάθος θα έχουν την δυνατότητα να το κάνουν αυτό στις 4 Σεπτεμβρίου όπως μόλις μα ενημέρωσε ο εισηγητή, και στις 11 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. 8 Οκτωβρίου θα εξετήσουμε τι τροπολογίε. Ε, στην... Θα συζητήσουμε το θέμα στις 5 Νοεμβρίου εδώ στην ΕΚΟΝ και στη συνέχεια θα πάει στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν που ε, ακολουθείτε αυτό το σφιχτό πρόγραμμα και Τώρα έχουμε ένα 25 λεπτό διάλειμμα πρωτού επανέλθουμε εδώ και μετά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό θα περάσουμε στις 12 και 4 στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ.